Uh, Γεια σας παρακαλώ. Να καθίσετε παρακαλώ. Καταρχάς κηρύσω την έναρξη φυσικά της συνεδρίασης αυτής και να σας ζητήσω αν κάνετε δεκτή την ημερήσια διάταξη. Πρέπει να εγκρίνουμε επίσης τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 14ης Απριλίου, 1ης και 2ης Ιουνίου και 28ης Ιουνίου. Δεν έχουμε σχόλια και από την αυτή την κατάσταση στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν έχω ανακοινώσεις. Then we have to do point which is the... Και το 4 είναι η αποδοχή του χρονοδιαγράμματος συνεδριάσεων για το 2011. Έχει γίνει μία πρόταση, δεκτή έγινε από τους συντονιστές την 6η Σεπτεμβρίου. Εν πάση περιπτώσει πριν το τέλος της συνεδρίασης, αν έχετε παρατηρήσεις να τις κάνετε, γιατί αλλιώς θα θεωρήσουμε φυσιολογικά ότι η πρόταση των συντονιστών γίνεται δεκτή. Περνάω ήδη στο σημείο 5. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω τον Ζαν Τρισσέ, τον πρόεδρο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Από τον, Ιούλιο έχουμε, από τον Ιούνιο έχουμε να τα πούμε. Θα έχουμε άλλη μια συνάντηση στις 30 Νοεμβρίου. Είναι τακτικός επισκέπτης μας βέβαια ο κύριος Τρισέ και θα ήθελα να τον καλωσορίσω. Ο κύριος ε, Τρισέ θα μας μιλήσει περίπου για 15 λεπτά, θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες οικονομικές και χρηματοπιστές ε, εξελίξεις. Θα μας μιλήσει επίσης και για θέματα φορολογικών πολιτικών. Θα είναι τμήμα της ευρύτερης συζήτησης. Θα ζητήσουμε επίσης και τα θέματα της μορφής της οικονομικής διακυβέρνησης και της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, 1,5 λεπτό ο καθένας και 3,5 λεπτά για τον Πρόεδρο για να απαντήσει. Θα ήθελα να πω ότι μέσα στο 1,5 λεπτό θα πρέπει να θέσετε μία ερώτηση παρακαλώ. Δεν είναι καθόλου ευγενές να ζητήσει κανείς ε, μια πλήρη απάντηση σε 10 ερωτήσεις τις οποίες θα θέσετε σε τόσο μικρό ε, χρονικό διάστημα. Κύριε Τρισέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, Πρόκειται για την τακτή θα έλεγα συνάντηση την εποχή που υπάρχει σημαντική πρόοδο στην Ευρώπη σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή σας για την υιοθέτηση του πακέτου χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Βλέπω πόσο το Κοινοβούλιο εργάστηκε στα θέματα αυτά σκληρά και αυτό μου δείχνει ότι το θεσμικό αυτό όργανο έκανε ένα τεράστιο ποιοτικό άλμα για να αποκτήσει το ρόλο τον οποίο του αποδίδει η συνθήκη της Λισαβόνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βοηθήσει για να υιοθετηθεί μια πολύ φιλόδοξη ημερήσια διάταξη για μεταρρυθμίσεις με μια πραγματικά ευρωπαϊκή προοπτική. Σαν θεσμικό όργανο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εντυπωσιαστεί τα μάλα από τις προσπάθειές σας και την στήριξή σας. Ένα άλλο νομοθετικό πακέτο, συνεχίζει γαλλικά ο Πρόεδρος, θα συζητηθεί ε, αυτή την εβδομάδα. Η μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ικανότητα και επίσης την επιθυμία του Κοινοβουλίου και της δικής σας Επιτροπής να επιδιώξετε για μια ακόμη φορά μια ευρωπαϊκή άποψη γύρω από την υπόθεση αυτή. Και εδώ έχουμε ανάγκη από ένα ουσιαστικό ποιοτικό άλμα για να διασφαλίσουμε μια καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς των 27 χωρών και μιας πλήρους συνοχής της νομισματικής ένωσης που είναι ο πυρήνας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. συνήθως ε, και σήμερα θα αναφερθώ στις ε, αξιολογήσεις, στις προβλέψεις ε, της ε, τράπεζας όσον αφορά στην τρέχουσα κατάσταση. Και κατόπιν θα ήθελα να αναφερθώ, να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο θέματα. Αφενός στη μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου θα αναφερθώ στο μέλλον της ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς ρύθμισης χρηματοπιστωτικών αγορών. Να περάσω τώρα στα θέματα των εξελίξεων στον οικονομικό και νομισματικό τομέα. Μετά από την τελευταία συνάντηση που είχαμε τον Ιούνιο, τα πράγματα στα, στις, στα στοιχεία τα οποία έχουμε λάβει πάνε καλύτερα από ό,τι νομίζαμε έχουμε μια ανάπτυξη της οικονομίας κατά 1% περίπου ανατρίμηνο, συνολικά στο τέλος του χρόνου θα φτάσουμε στο 4%. Πιστεύουμε ότι ακόμα παραπέρα θα συνεχιστεί αυτή η ήρεμη θα έλεγα μορφή ανάκαμψης της οικονομίας, αλλά με μια σαφέστατη υποβόσκουσα εν πολλής όθηση η οποία θα βελτιώσει την κατάσταση παρά τις αβεβαιότητες που υπάρχουν. Ο πληθωρισμός είναι 1,6 τον Αύγουστο, ε, υπάρχει μια μικρή μείωση από το 1,7 του Ιουλίου όπως προεβλέπεται. Στο μέλλον πιστεύουμε ότι ο ρυθμός της ανάπτυξης βαχυπρόθεσμα θα αυξηθεί, αλλά θα πρέπει να παραμείνει, θα έλεγα, σχετικά χαμηλά σύμφωνα με τις προβλέψεις σε συγκεκριμένους τομείς. Νομίζω ότι οι προσδοκίες στον τομέα του πληθωρισμού είναι πάντα στα πλαίσια τα οποία έχουμε ορίσει σύμφωνα με τον ορισμό τον οποίο δίδουμε στη σταθερότητα των τιμών. Η νομισματική ανάλυση την οποία κάνουμε επιβεβαιεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ελεγχόμενες. Αυτό φαίνεται και στους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της πίστοσης και του χρήματος, αύξησης μάλλον της πίστοσης και του χρήματος αυτή η χαμηλή και ελεγχόμενη ανάπτυξη και στη δανειοδοτική δραστηριότητα δείχνει ότι ε, η κατάσταση βελτιώνεται για τα νοικοκυριά, αλλά είναι αρνητική για τις επιχειρήσεις. Εμείς στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων τα οποία έχουμε αλάβει, συνεχίζουμε να επαναχρηματοδοτούμε ε, σε διαδικασίες μάλλον με σταθερά επιτόκια, και ελπίζουμε επίσης ε, να συνεχίσουμε τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στον τομέα των τραπεζών ε, χρηματοδοτώντας εκ νέου εξάμηνες και δωδεκάμηνες δραστηριότητες όταν αυτές οριμάσουν. Μέσω έτσι και αλλιώς του προγράμματος αγορών χρεογράφων συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε σε ε, ελεγχόμενα όμως επίπεδα σε ορισμένους τομείς της Ευρωζώνης στον τομέα των ομολόγων. Αυτή η παρέμβαση έχει σαν στόχο την βελτίωση της λειτουργίας της ε, νομισματικής μας πολιτικής. Συνολικά η ηγεσία της τράπεζας θεωρεί ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα και οι παρούσες συνθήκες είναι θα έλεγα εύθετες και δίνουν δυνατότητες οι οποίες είχαν προβλεφθεί και νομίζω ότι και το ύψος των επιτοκίων που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι τα κατάλληλα. Όλα τα μη τακτά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από το ευρωσύστημα σε εισαγωγικά κατά τη διάρκεια της ε, της έντασης που είχε δημιουργηθεί στις οικονομικές αγορές είναι συμβατά με τις βασικές μας πολιτικές απόψεις και δεν έχουν επηρεαστεί αρνητικά. Σχετικά με τις δημοσιονομικές πολιτικές, η επιστροφή σε αξιόπιστες, υγιείς φορολογικές πολιτικές είναι απαραίτητη. Γι' αυτό απευθύνουμε, θα έλεγα, έκκληση σε όλες τις χώρες να προχωρήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση κάποιες θετικές εξελίξεις στις ισροές φορολογικών εσόδων που μπορεί να υπάρξουν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά. Θα ήθελα να ασχοληθώ τώρα με συγκεκριμένα θέματα, ξεκινώντας με τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Ο πρόεδρος Φων Ρόμπαϊ σας ενημέρωσε πρόσφατα για τα βήματα προόδου τα οποία έγιναν από την Task Force της οποίας προεδρεύει. Προπόησε σε ορισμένα σημεία, ιδίως του Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Σε άλλα ζητήματα όπω την ενισχυμένη δημοσιονομική εποπτεία και, μια νέα, και ένα νέο πλαίσιο μακρονομική εποπτεία, χρειάζεται περισσότερη φιλοδοξία και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις κυβερνήσει του ζώνης ευρώ κεντρικός στόχο θα πρέπει να είναι να πετύχουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τη νομισματική μα Ένωση. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει την ε, ε, Τι ε, νομοθετικέ της προτάσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω σύνομοθετή, θα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού ενός αποτελεσματικού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσει για το εποπτικό πακέτο έδειξαν ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι πρόθυμο να δεχθεί συμβιβασμού στη βάση του ελάχιστου κοινού παρανομαστή. Ιδεοδός, για να έχουμε ένα ποιοτικό άλμα στην ενίσχυση τη οικονομική διακυβέρνηση τη Ένωση και τη ζώνη του ευρώ θα χρειαζόταν αλλαγή τη συνθήκη. Αυτό σημαίνει ότι οι χώροι, εφόσον δεν υπάρξει μια τέτοια ταχεία και η άμεση αλλαγή τη συνθήκη, πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυνατό όλε τι δυνατότητε τη παράγωγης νομοθεσίας της Ένωσης με την φυστάμενη ε, συνθήκη να πετύχουμε αυτό το ποιοτικό άλμα. Η τράπεζα υπολογίζει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου στην πίστη τη ότι ο δεδομένη μεταρρύθμιση τη οικονομική διακυβέρνηση ιδίω τη ζώνη του ευρώ χρειάζεται για να εκμεταλλευτούμε πλήρω τι δυνατότητε που προσφέρει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Το μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Τράπεζα, κ. Μπίνη Μάγκη, σα παρουσίασε πρόσφατα τη θέση μα για, βα... για διάφορες πτυχές τη οικονομική της μεταξύ των οποίων μια σειρά θεμάτων που αφορούν την επίλυση κρίσεων. Επίσης υπογράμμισε την οικονομική λογική που στηρίζει τη θέση μας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που εμείς θεωρούμε απαραίτητα στοιχεία για ένα μεταρρυθμισμένο πλαίσιο δημοσιονομικής και μακροοικονομικής εποπτείας που είναι στο κέντρο των ε, τρεχουσών συζητήσεων. Το νέο πλαίσιο θα έπρεπε να έχει σωστό να είναι σωστά το στοχοθετημένο, ιδίω σε χώρε με υψηλό χρέο και μεγάλε απώλειες ανταγωνιστικότητας. Το επίπεδο του δημοσίου χρέου και εξέλιξη των ελλημάτων μπορεί να είναι πηγή ε, ε, χρηματοοικονομικής αστάθειας και να μεταδοθούν σε άλλες χώρες με το ίδιο νόμισμα. Άρα το χρέος θα έπρεπε να έχει ενισχυμένο καθεστώς στην δημοσιονομική εποπτεία, τόσο στο σκέλος πρόληψης, όσο και στο σκέλος διόρθωσης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η προοδευτική απώλεια, η απώλεια ε, ανταγωνιστικότητα στην νομισματική ένωση αποτελούν άλλη πηγή ακραία αστάθεια. Ένα νέο σύστημα εποπτείας για τον έλεγχο και διόρθωση των μακροοικονομικών ασταθειών όπου ανακύπτουν χρειάζεται κατά συνέπεια. Η ιδέα αυτή απέκτησε αρκετή υποστήριξη αλλά χρειάζεται να συμφωνηθούν συγκεκριμένα μέτρα για να καταστεί λειτουργική και παρκώς δεσμευτική. Όταν εντοπίσουμε τις αβεβαιότητες και τα τροτά στοιχεία, πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική συνέχεια και συγκεκριμένες αποστολές αναχώρα, ειδικέ συστάσεις πολιτικής, αύξηση ε, δημόσιας πίεσης από άλλα κράτη και εν τέλει ένα ε, πλέγμα σαφών μέτρων διόρθωση. Εφόσον τα τροτά στοιχεία σε κάποιο μέρο μπορεί να έχει συνέπειε, άμεση συνέπειε σε άλλο μέλο, το πλαίσιο εποπτεία θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα κλιμακούμενο σύστημα κινήτρων και ε, κυρώσεων που μπορεί να ενεργοποιηθεί επαρκώ έγκαιρα στη διαδικασία και μπορεί να λειτουργεί κατά τη στοιχεία με το βαθμό της παράπτωσης. Και μάλιστα ένα βασικό απαραίτητο κύριο στοιχείο αποτελεσματικού μηχανισμού εποπτείας είναι ένας λειτουργικός μηχανισμός κινήτων και κυρώσεων και χρηματοοικονομικού και μη χαρακτήρα, ιδίως για τις χώρες της νομισματικής ένωσης. Είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει ένα μια φιλόδοξη θέση στο ζήτημα αυτό. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι σχεδόν αυτόματες βάσει προτάσεων της Επιτροπής και όχι συστάσεών της. Η Τράπεζα πρότεινε αντιστροφή των διαδικασιών ψηφοφορίας που οδηγούν στην οθέτηση των κινήτων και των κυρώσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί εκτός αν η ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο καταψηφίσει την πρόταση της Επιτροπής. Ο ρόλος λοιπόν της επιτροπή κατά συνέπεια θα αυξηθεί σημαντικά. Επιπλέον, για να ενσωματώσουμε τις απαιτήσει συμμετοχή στην Νομισματική Ένωση, ε, οι ευρωπαϊκοί κανόνες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί και να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη με ισχυρά εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια και τη δημιουργία ανεξάρτητων ισχυρών ε, θεσμών παρακολούθησης και υιοθέτηση εθνικών φορολογικών κανόνων που θα αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις, θα τις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία της εξέλιξης. Βάσει των ε, ζητούμε να ενισχυθούν οι υποχρεώσεις και εξουσίες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και να ενισχυθούν οι εντολές συλλογής στοιχείων ακρίβειας των πόρων ακρίβειας και ακρίβειας του ελέγχου. Οι αλλαγές θα πρέπει να ξεπεράσουν τον πρόσφατο κανονισμό για τη Eurostat. Αυτό που είναι επίσης κρίσιμο είναι η ανεξαρτησία της ανάλυσης, της κρίσης και της ε, παρακολούθησης που δεν πρέπει ποτέ να τεθούν ξανά υπό αμφισβήτηση. Περιμένω από την Επιτροπή να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις για, τη μεταρρύθμιση διακυβέρνησης στους τομείς αυτούς για να ενισχυθεί η ανεξάρτητη δημοσιονομική παρακολούθηση, η Τράπεζα θεωρεί ότι είναι καλό να υπάρχει μια συμβουλευτική δομή ε, σοφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα παρέχει δεύτερη άποψη. Συνοπτικά, ο κατάλογος της αναθεώρησης των προτάσεων για την διακυβέρνηση της ζώνης ευρώ θα πρέπει να είναι θετικές απαντήσεις στα επόμενα πέντε ερωτήματα. Πρώτον, η το πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες, σωστά καλύπτει τις αδυναμίες που, που προέκυψαν για να αποφευθεί νέα κρίση. Δεύτερον, χρειάζεται αυτή η εποπτεία να λειτουργεί δυνατότητα, να, να ξεκινά δυνατότητες προσαρμογής ε, ε, ανισοτήτων. Τρίτον, οι μηχανισμοί εφαρμογή και υλοποίηση τη ε, της είναι σχεδόν αυτόματοι και ε, οι κυρώσει μπορούν να προστατεύσουν τα άλλα μέλη και την νομισματική ένωση. Τέταρτον, το πλαίσιο περιλαμβάνει επαρκή ανεξαρτησία και εποπτεία και απαραίτητα στοιχεία ελέγχου τη ποιότητα, τη ανάλυση των στατιστικών. Και τελευταίο σημείο. Οι νέε αρχέ οικονομική διακυβέρνηση συνδέονται με το εθνικό πλαίσιο. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στι επόμενε μέρε τι απαντήσει στα ερωτήματα αυτά που έδωσε η ομάδα εργασία υπό τον κύριο Βάνερον και το Κολέγιο των Επιτρόπων από την άλλη πλευρά και ελπίζω να μπορέσουμε να καλύψουμε τις κρίσιμες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Αν, είναι, οι απαντήσει αν αυτές είναι δειλές κατά την απόψή μας, θα, θα προσέλθουμε ενώπιον σας και θα το πούμε. Να αναφερθώ τώρα στη, στα κάποια επερχόμενα ζητήματα. Πολιτικό momentum αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την ε, ε, γενικότερη ενίσχυση της κανονιστικής προσέγγισης. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το δυναμισμό και να τον διατηρήσουμε. Η Βασιλεία δύο είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, διότι αποτελεί τον πυρήνα των ε, δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και επιφέρει την ισορροπία ανάμεσα στον ευρύτερο στόχο που είναι η ενίσχυση της αντίστασης του χρηματοπιστωτικού τομέα και της ανάγκης στήριξης ε, δανειοδότησης και χορήγηση δανείων στην πραγματική οικονομία. Βεβαίως ε, δεν μπορώ να μιλήσω για την εποπτεία χωρίς για άλλη μια φορά να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έγκριση του πακέτου μεταρρύθμισης τη εποπτείας. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κινδύνου και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή από κοινού ε, θεωρώ ότι θα καταστήσουν το πλαίσιο πιο ανθεκτικό και θα δώσουν δυνατότητα σε όσους ασκούν την εποπτεία και τη ρύθμιση να καθορίσουν, να καθοδηγήσουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσα από μια πραγματική οικονομία η οποία θα αντέχει τις ε, προκλήσεις ε, και θα μπορέσει να αποφύγει τις υπερβολές και τα πλεονάσματα καθώς λοιπόν περνάνε οι κρίσιμες περίοδοι εμείς ε, θεωρούμε ότι ο νέος αυτός φορέας θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το νέο λοιπόν αυτό οικοδόμημα των ε, μεταρρυθμίσεων και της ρύθμισης είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολούν. Υπάρχει και οδηγία για, τα εναλλακτικά, για τις εναλλακτικές απενδύσεις που είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ένα εναλλακτικό εργαλείο επενδύσεων. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σωστό να υπάρχει έγκαιρη αναφορά στις αρχές που ασχολούνται με τις επενδύσεις, ε, όπως επίσης και να ελέγχουμε τους συστημικούς κινδύνους. Υπάρχει πρόοδο στην νομοθεσία για τις ακάλυπτες πωλήσει. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των ρυθμίσεων. Τέλος, ε, ε, υπάρχουν συστημικοί σημαντικοί θεσμοί που πρέπει να ελέγχονται. Το πρόβλημα των αρνητικών κινήτρων που απορρέει από υπερβολική εξάρτηση από εξωτερικές αξιολογήσεις και αυτό το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή της μεταρρύθμισης, θα είναι μια μακρά διαδικασία και θεωρώ ότι οι αρμόδιες αρχές θα επιδιώξουν να επιτύχουν τους στόχους μας, στόχους που οι πολίτες θεωρούν ότι είναι απολύτως απαραίτητοι και θα προκύψει μέσα από άοκνες προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε λοιπόν στη σειρά των ερωτήσεων. Όχι πάνω από 1,5 λεπτό. Όχι πολλαπλές και περίπλοκες ερωτήσεις. Ο κύριος Γκοζές είναι ο πρώτος εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα μοιράσω τη σειρά γενικά των παρεμβάσεων ανάλογα με τις πολιτικές ομάδες. Κύριος Γκοζές, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, θα ήθελα να συγχαρώ τον μελλοντικό Πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικών Κινδύνων. Το Κοινοβούλιο πράγματι ε, θέλησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας, λόγω ακριβώς της ιδιότητάς του αυτής, να αναλάβει Πρόεδρος της συγκεκριμένης Επιτροπής. Ελπίζω την επομένη φορά να μας πείτε για την οδηγία για το Δέλτα Νιτάφ, αυτά που μας είπατε για την εποπτεία. Ότι έφτασε η εποπτεία δηλαδή έγκαιρα και δίνει ενδιαφέρουσες λύσεις. Οι διαπραγματεύσεις ε, για την οδηγία αυτή συνεχίζονται και είναι σκληρές ε, διαπραγματεύσεις γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να βάλει μια νότα Ευρώπης σε αυτές τις ε, οδηγίες και τις ρυθμίσεις και τι σχόλια μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να καταλάβουμε πώς θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος Τρισέ. Θα ήθελα να εκφράσω για μια ακόμη φορά την εκτίμησή μου στην τεράστια προσπάθεια που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας τους τελευταίους μήνες και στα πλαίσια της οδηγίας αυτής. Έχει μεγάλη σημασία η οδηγία αυτή γιατί θα έλεγα αντιμετωπίζει ένα θέμα το οποίο δεν είναι τόσο απλό και ξεκάθαρο όσο κάποια άλλα θέματα όπως σαν παράδειγμα η εποπτεία των τραπεζών σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας της αγορός, το θέμα των λεγόμενων highly leveraged institutions, Αυτό το οποίο έχει σημασία στην Ευρώπη είναι να υπάρξει ένα σύστημα εποπτείας, ένα σύστημα διαφάνειας, το οποίο να είναι το καλύτερο στον κόσμο ή στο καλύτερο επίπεδο στον κόσμο. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μην υπάρχουν διαφορές εδώ ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί η αδίποτε μορφή διαφοράς θα, θέσει, θα δημιουργήσει προβλήματα, ε, μίζωνα προβλήματα, διεθνούς αστάθειας η οποία θα παραμένει γιατί οι διάφοροι χρήστες θα μετακινούνται προς τις περιοχές τις οποίες θα υπάρχει ο μικρότερος διακανονισμός. Οπότε η διακανονιστική διαιτησία θα έλεγα, η επιλογή θα λειτουργήσει αρνητικά για τη διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα υπάρχουν μετακινήσεις δραστηριοτήτων αναπόφευκτα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε σε συνεργασία με τους Αμερικανούς να έχουμε ένα δίκαιο πεδίο θα έλεγα το οποίο θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που είναι πάντα απαραίτητη. Ως προς αυτό να σας πω ότι είναι προφανές ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Είναι απαραίτητο αυτό. Είναι επίσης απαραίτητο, είναι προφανές μάλλον, ότι και σε επίπεδο αρχών και σε επίπεδο ακαδημαϊκών χώρων, πανεπιστημίων κτλ. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα στοιχεία ε, που προκαλούν συστημικές αστάθειες. Αυτά τα στοιχεία θα έλεγα δημιουργούν φοβίες σχετικά με τη λειτουργία αυτών των οργανισμών. Ως εκ τούτου ε, και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπεζά αλλά και για το σύνολο των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών αλλά και το σύνολο των ερευνητών πανεπιστημίων κτλ. Είναι ένα τομέας στον οποίο πρέπει να δουλέψουμε πολύ ακόμα για να μπορέσουμε να πιστέψουμε ότι θα κατανοήσουμε τις συστημικές αστάθειες οι οποίες συνοδεύουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ευχαριστώ, Πριν από δύο περίπου εβδομάδες ε, σας συναντήσαμε στη Φραγκφούρτη και εκεί είχα την ευκαιρία η διεισόμαση να διαπιστώσω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, εργάζεται πυρετοδός για την νέα ρυθμιστική αρχή, την ευρωπαϊκή. Πιστεύετε ότι θα έχετε ολοκληρώσει προσπάθειές σας έγκαιρα και θα μπορέσει να λειτουργήσει η ρυθμιστική αυτή αρχή την πρώτη πρώτου του επόμενης χρονιάς. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής. Εμείς οι βουλευτές τα τελευταία χρόνια επισημαίνουμε ότι η ευρωπαϊκή οικονομική η Ευρωζώνη δεν είναι ισορροπημένη. Δηλαδή ένα κοινό νόμισμα μπορεί να λειτουργεί σωστά μόνο εφόσον υπάρχει και συνεργασία και αρμονία στις ε, οικονομικές ε, και ε, χρηματοπιστωτικές πολιτικές των κρατών μελών. Χαιρόμαστε που το αναγνώρισαν αυτό και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Όμως ακόμα δεν έχουν ρυθμιστεί όλε τι λεπτομέρειες. Γι' αυτό λοιπόν εν ώψη της συνάντησης κορυφής θα μπορέσετε εσεί να αποχωρήσετε αυτό το σχέδιο και ή δυνατόν εξ εξισορροπήσετε και τις ε, ανομαλίες και ανισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. On your first question. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, ε, νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και βεβαίως ε, αυτό το κάνουμε ευθύς εξ αρχής. Υπάρχει αυτή η ιδέα του Systemic Risk Board, του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, Αντιμετωπίσεων Συστημικού Κινδύνου, συστημικών κινδύνων που ε, θα τεθεί σε λειτουργία, θα αρχίσει να λειτουργεί από την 1η Πρώτου του 2011. Είμαστε σε επαφή με τους ε, διοικητές ε, των 27 κρατών μελών, με το Γενικό Συμβούλιο. Βεβαίως οι ευθύνες που φέρουμε είναι πολλές και θα δούμε όταν ε, θα υπάρχει αυτό το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα δούμε πώς θα ε, οργανώσουμε τη δουλειά μας. Πάντως ε, θα υπάρχουν τα εργαλεία, θα υπάρχει ο εξοπλισμός. Οφείλω βέβαια να αφήσω κάποιο περιθώριο και στον ίδιο τον φορέα, στην ίδια την αρχή, γιατί όπως και εσείς σωστά είπατε, μόνοι τους θα πρέπει να δρομολογήσουν τη δουλειά τους. Είναι δηλαδή δυνατόν στην αρχή, η αρχή αυτή να μην είναι απόλυτα λειτουργική, αλλά παρόλα αυτά, αν μου επιτρέπετε να πω, η επικεφαλής των ευρωπαϊκών ομάδων που φέρουν σήμερα την ευθύνη για την εποπτεία των ε, τραπεζών, των ε, αγορών, αυτοί θα υπάρχουν, θα αρχίσουν να λειτουργούν ευθύ εξ αρχή. Ίσως, σε πάση περιπτώσει, χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο, που βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτα δική μα ευθύνη. Αλλά όσον αφορά το ESRB, το ε, Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων, είμαι αρκετά αισιόδοξο. Θέλω επίση να πω το εξή. Κατά τη δική μου γνώμη, σε αυτόν τον τομέα της ε, εποπτείας δημοσιονομικών πολιτικών, υγιών δημοσιονομικών πολιτικών, που πρέπει να εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις, εμείς, κατά τη δική μου πάντα άποψη, δεν μπορούμε να επιτύχουμε το βέλτιστο, γιατί υπάρχει μία μόνιμη υποτίμηση του τι είναι απαραίτητο να λάβει χώρα σε αυτό τον τομέα. Το μήνυμά μας είναι το ίδιο. Γνωρίζετε ότι κατά το παρελθόν υπήρξε μία ε, ιδιόμορφη υποτίμηση της κατάστασης. Το 2004, το 2005 αναγκαστήκαμε να διαφυλάξουμε και να επιβάλλουμε το σύμφωνο σταθερότητας που τότε κρίθηκε ως μια παράλογη, ένας παράλογος περιορισμός ε, των δημοσιο... στις δημοσιονομικές πολιτικές. Βλέπετε λοιπόν τι έγινε και όλοι γνωρίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό να τηρείται αυτή η πολιτική. Το είπα εξάλλου στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις ότι εμείς θα συνεχίσουμε να καλούμε όλες τις κυβερνήσεις να εργάζονται όπως αναμένεται. Πρέπει βέβαια να πω ότι υπάρχει ένα θέμα διακυβέρνησης ε, που αυτή τη στιγμή διακυβεύεται και αναμφίβολα θα είμαστε σε επαφή στο μέλλον γιατί και εσείς ε, έχετε μεγάλη ευθύνη σε αυτό το θέμα της ε, νέας μορφής διακυβέρνησης. Χωσέ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για τις συζητήσεις που είχαμε για το Συμβούλιο Συστημικών Κινδύμων μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής, αλλά και ημών. Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση με σαφήνεια. Στο θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας, το σύμφωνο σταθερότητας και τις κυρώσεις ιδίω, πέραν των τις οικονομικές κυρώσεις, όχι τις πολιτικές, οι ερωτήσεις είναι σαφείς. Πιστεύετε εσείς, εσείς ως πρόεδρος, οι κυρώσεις πρέπει να είναι αυτόματες ή να εξαρτώνται από αποφάσεις του Συμβουλίου. Έχει νόημα αυτή τη στιγμή να διατηρήσουμε διαφοροποιημένες κυρώσεις για τις χώρες της ζώνης ευρώ από τις χώρες που είναι εκτός. Τρίτον, οι κυρώσεις, οι οικονομικές κυρώσεις πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία με τόσο στην, στα προβλήματα ελλείμματος όσο και στα προβλήματα χρέους ως μη τήρηση της αρχής της, ε, ε, θεωρείται ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα στην αρχή της ε, μη, ε, της μη ανταγωνιστικότητας που είναι βασική αρχή της συνθήκης. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως είπατε, Ε, στον τομέα των κυρώσεων υπάρχουν κάποιες κυρώσεις που μπορεί να είναι ε, απολύτως εύκολα λειτουργικές στα πλαίσια της υφιστάμενης συνθήκης και χρησιμοποιώντας όλη την παράγωγη νομοθεσία και άλλες που να είναι δυσκολότερες. Εξετάζεται, είναι ακόμα υπό εξέταση κατά πόσον οι πολιτικές κυρώσεις, αναστολή δικαιώματος ψήφου κλπ. μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή όχι. Εμείς θα υποστηρίζαμε κάτι τέτοιο, διότι είναι κάτι που δεν είναι οικονομική, χρηματοοικονομική κύρωση, αλλά έχει μεγάλο αντίκτυπο, μεγάλη, πολλές συνέπειες. Είναι ωστόσο ενδεχόμενο να, χρειαστεί, να χρειαστεί κάτι τέτοιο αλλαγή συνθήκης. Η δική μας αντίληψη ωστόσο είναι η εξής. το να έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα χωρίς να έχουμε μια πολιτική ομοσπονδία και το έλεγα αυτό εδώ και πολλά χρόνια λειτουργήσαμε παράτολμα δεν έχουμε πολιτική ομοσπονδία έχουμε ενιαίο νόμισμα πρέπει να αποκτήσουμε το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για τον έλεγχο και την ενίσχυση της εποπτείας όχι μόνο στο, δημοσιο... φορολογικό πλαίσιο, στο δημοσιονομικό συγγνώμη πλαίσιο, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο όσο καλύτερα γίνεται, θα έλεγα αυτό θα επιτευχθεί όχι μόνο με την ιονή αυτοματικότητα, αλλά και με την αντιστροφή της διαδικασίας. Περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις και θα κρίνουμε εμείς. Θεωρούμε ωστόσο ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ μακριά με την υφιστάμενη παράγωγη νομοθεσία χωρίς να αλλάξουμε αμέσως τη συνθήκη. Για την τελευταία ερώτησή σας, ε, ε, έλλειμμα και χρέος. Είναι σαφές ότι αυτό που μετράει για τους εξωτερικούς παρατηρητές, για τους επιχειρηματίες, για τους επενδυτές, για τους αποτιμιευτές, είναι ο συνδυασμός εκρεμούς χρέους και ελλείμματος. Αυτό επιτρέπει σε κάποιον να ελέγξει και το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και να μειώσει επαρκώς γρήγορα το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ για να αποκτηθεί η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό θεωρούμε ότι μέχρι τώρα τα κριτήρια του χρέους είχαν παραμεριστεί, είχαν ξεχαστεί. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να στηριχθούμε και στις δύο και πρέπει να εξετάζουμε και τα δύο, όπως το λέει άλλωστε και τα κριτήρια του Μάστεχτ. Μαζί και έλλειμμα και χρέος, διότι είναι θεμελιώδες για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη ξανά, να αποκαταστήσεις την κατάσταση. Ευχαριστώ. Περβάνς. Κύριε Πρόεδρε, μας είπατε ότι σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσουμε σε μια πρώτη φάση θετικά σε πέντε ερωτήσεις. Υπάρχει μια ερώτηση όμως την οποία δεν αναφέρεται. Η ερώτηση είναι το τι θα γίνει με τον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων έτσι όπως διαμορφώθηκε αυτός ο μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με την ελληνική περίπτωση που κατέστησε εύθραυστη εν πολλής ε, την ζώνη ευρώ. Μπορούμε λοιπόν να, χρησιμοποιήσουμε αυτό το ισχυρό μέσο το οποίο δημιουργήσαμε και το οποίο βέβαια θα πρέπει να αποκτήσει μια κάποια χρονική διάρκεια. Και αυτή η διάρκεια θα οδηγήσει να de devenir aussi attractif que le marché euh, américain à un Έχει ενδιαφέρον να βλέπει κανείς ότι κάποια ταμεία διεθνή ε, τα οποία εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την Αμερικανική αγορά παρότι είναι η αγορά η οποία γέννησε τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και βλέπουμε και ευρωπαϊκές χώρες από την άλλη να δυσκολεύονται πολύ να χρηματοδοτηθούν από τη διεθνή αγορά κεφαλαίων. Ε, ε, όπως είπα, υπήρξε εδώ ένα μέλος του Δικητικού Συμβουλίου που έδωσε αρκετές απαντήσεις σχετικά με το μηχανισμό κρίσης και με την χρηματοπιστωτική σταθεροποίηση σε εποχές κρίσης. Και θα ήθελα να συγκεντρώσω και εγώ την προσοχή μου σε αυτά τα οποία πρέπει να αποφύγει κανείς για να μην τύχει σε μια τέτοια κατάσταση. Συγγνώμη, διακόπτη κυρία Πέρες. Η ενσωμάτωση του χρέους δεν είναι μηχανισμός αντιμετώπισης της κρίσης. Κοιτάξτε, εγώ απαντώ στο πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο τώρα σχετικά με την ενσωμάτωση του χρέους. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν σαφής. Θεωρούμε ότι τα διάφορα λογιστήρια και οι διάφορες εθνικές κυβερνήσεις έχουν τις δικές τους ευθύνες. Και αυτό δεν είναι καθόλου κακό είναι υπεύθυνε για τις πολιτικές που ακολουθούν. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό το οποίο μας έλειψε είναι κάποια κίνητρα έτσι ώστε να υπάρξει μια εθνική, εσωτερική αν θέλετε, σωστή διαχείριση. Αυτό μας έλειψε. Εγώ εξέφρασα την απογοήτευσή μου για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η εποπτεία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης πάρα πολύ μέτρια τα πράγματα και από όλου τους εμπλεκομένους δεν υπήρξε η αίσθηση ότι υπήρχε μια πραγματική επιθυμία να υπάρχει ένας αμοιβαίος σε εισαγωγικά έλεγχος. Ξέρετε ότι σε κάποια φάση οι κυβερνήσει θέλησαν αυτή η αμοιβαία επίβλεψη και εποπτεία να διαλυθεί πλήρως. Πέραν αυτού και επιπλέον των μέτρων τα οποία προβλέπουμε να ληφθούν και απαντούμε και προσδοκούμε θετικές απαντήσεις και στις πέντε αυτές ερωτήσεις, ένας μηχανισμός διαχείρισης κρίσης είναι σίγουρα δυστυχώς απαραίτητος και ελπίζω ότι στο μέλλον η αποφασιστικότητα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου φυσικά και κυρίως τα μαθήματα της εμπειρίας την οποία βιώνουμε την εποχή αυτή, η οποία είναι μια πολύ δύσκολη αντικειμενικά περίοδος, θα μας επιτρέψουν με εξαιρετικό τρόπο να θωρακίσουμε τα μέσα εποπτείας μας, που θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε στο μέλλον καταστάσεις σαν και αυτές τις οποίες βιώσαμε. Ο κύριος Μπέρμαν. Κύριε, στη Γαλλία είναι υπεύθυνο τη αρχή εποπτεία των χρηματοοικονομικών αγορών ανέφεραν ότι, χρημα... ότι χρησιμοποιήθηκε από τι αγορέ η κρίση στην Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκε, εκμετάλλευση. Χαιρόμαστε που ψηφίσαμε πρόσφατα μια δομή ευρωπαϊκή εποπτεία. Πιστεύετε ότι αυτέ οι δομέ θα έχουν επαρκή μέσα για να αποκαλύψουν μια τέτοια μελλοντική εκμετάλλευση, χρησιμοποίηση. Και τι θα χρειαζόταν για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Το υπάρχει επαρκής ε, νομικό οπλοστάσιο και επειδή κάτι τέτοιο το βρίσκει κανείς στο τέλος, ο ρόλος της τράπεζας είναι ουσιαστικός για να, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια καταχρηστική εκμετάλλευση και αντιμετώπιση της κατάστασης. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια όρια. Ποια είναι αυτά. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις ακάλυπτες πωλήσει στο short selling. Έχετε κάποιο σχόλιο με μια σειρά νομοθετικών κειμένων. Έχετε κάποιο σχόλιο. Μήπως θα έπρεπε απλά και μόνο να απαγορευτούν ορισμένα παράγωγα προϊόντα στην Ευρώπη και αλλού. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Euh, euh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση. Ε, τα πράγματα είναι σαφή. Υπάρχουν συμπεριφορές που είναι σύνομες και άλλες που δεν είναι. Υπάρχουν πράξεις που επιτρέπονται και πράξεις που δεν επιτρέπονται. Και πρέπει να πω ότι σε κάποιο κράτος δικαίου πρέπει να είμαστε να απαιτούμε απόλυτα την διάκριση μεταξύ του επιτρεπόμενου και του μη. Τώρα, το αν έγινε αντικείμενο εκμετάλλευση ή όχι μία πράξη ή όχι, δεν μπορώ να σου το πω εγώ, αλλά αν έγινε κάτι τέτοιο ξεκινούν έρευνες και ε, υφίστανται κυρώσεις αυτοί που, έχουν διαπράξει τις πράξεις αυτές. Αυτό ισχύει στην Ευρώπη και ισχύει σε όλες τις αγορές την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι, ίδιες οι κεντρικές τράπεζες έχουν σημαντικές ευθύνες, έχουν τη δική τους οπτική, που είναι μια οπτική σταθερότητα τιμών μέσω και μακροπρόθεσμα, χρηματοοικονομικής σταθερότητας μέσω και μακροπρόθεσμα στο μέτρο που εξαρτώνται από την αρχική αυτή έννοια της σταθερότητας των τιμών και έχουν και πολύ σημαντικές ευθύνες διότι κατά ανάγκη λόγω της λειτουργίας τους αυτής καθευτής βλέπουν μακριά, όχι βράχη πρόθεσμα. Και είναι ανεξάρτητες, που σημαίνει ότι επιτρέπεται, μπορούν να κάνουν την πιο ενδεδειγμένη κρίση μπορούν, μπορεί ωστόσο να έχουν ή να μην έχουν ευθύνε προληπτική εποπτεία, τραπεζική ή άλλη, και να έχουν ευθύνε εποπτεία στον τομέα της, ε, των ασφαλιών ή αλλού. Δεν πρέπει λοιπόν να συγχαίουμε τα πράγματα. Και στην πρόσφατη νομοθεσία που επένεσα προηγουμένως, το European Board που δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων, δεν συγχαίει τη δική του λειτουργία με αυτή των εποπτικών αρχών αυτών καθεαυτών, οι οποίες θα έχουν τις δικές τους ευθύνες σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω λοιπόν εκ νεού ότι το ερώτημά σας απευθύνεται περισσότερο προς, αυτούς, προς αυτές τις εποπτικές αρχές, είτε τραπεζών, είτε ασφαλιστικών επιχειρήσεων αν έγιναν τα λάθη από ε, αυτές τις δομές, ή τους επόπτες των χρηματοοικονομικών αγορών αν οι ανομαλίες εμφανίστηκαν στις αγορές. Κάτι ακόμα για την πρώτη ερώτησή σας. Υπάρχει νομίζω συνένεση, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ως προς το εξής. Χρειάζεται να πηγαίνουμε πάντα προς την μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Αν υπάρχουν ζώνες αδιαφάνειας, Οπουδήποτε και να υπάρχουν μπορούμε να βρούμε τέτοιες συμπεριφορές. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να μας οδηγήσουν και το υπογραμμίζω αυτό στο να δώσουμε απαντήσεις που πρέπει να είναι πραγματικά παράλληλες απαντήσεις. Η δεμή θα είχαμε σε παγκόσμιο επίπεδο τις ίδιες ανισορροπίες, τα ίδια προβλήματα χρηματοοικονομικής αστάθειας και επιπλέον αυτή την ε, επιλογή νομοθεσίας, αυτό το αρμπιτράζ νομοθεσίας που θα οδηγεί σε ζώνες μικρού νομοθετικού, χαμηλού νομοθετικού πλαισίου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σε επίπεδο των, ε, του, του G20 και σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Thank you very Κύριε Τρισέ, είσαστε ε, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Συστημικών ε, Κινδύνων και θα ήθελα να σας ρωτήσω, ο στόχος της σταθερότητας των τιμών είναι συμβατός με το στόχο της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και με αυτή τη νέα σας ιδιότητα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου, αυτή η νέα ιδιότητα θα επηρεάσει την ε, νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης. Καταρχήν, να σας πω ότι ακόμα δεν είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Συστημικών Κινδύνων. Πρέπει να ακολουθήσει η νομική ε, διαδικασία. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Αυτό το ένα. Και κατά δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Συστημικών Κινδύνων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν αλλάζει τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων έχει τη δική της εντολή, έχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί και δεν αλλάζει τίποτα. Δεν θα αλλάξουν οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εσείς αναφερθήκατε στην Ευρωζώνη, άρα δηλαδή και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τιμικών Κινδύνων. Ήρθαν ε, παρόδο και ε, ξέρετε η σταθερότητα των τιμών είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα. 11,5 χρόνια είμαστε τώρα μετά την ε, ύπαρξη του ευρώ. Ο πληθωρισμός είναι ο μέσος 1,97% στην Ευρωζώνη. Και στην αρχή είχαμε πει κάτω από 2, κοντά στο 2. Είμαστε λοιπόν στο 1,97 ρυθμό πληθωρισμού, κάτω από το 2, κοντά στο 2. Άρα δηλαδή, τουλάχιστον σε επίπεδο αριθμών, είναι εντυπωσιακό. Θα μπορούσε ο πληθωρισμός να είναι 95 ή 1,90 εγώ προτιμώ το 97 από το 2,1, αν θέλετε να είμαι ειλικρινής. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος του έτους θα κάνουμε τους ακριβείς υπολογισμούς. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να πετύχουμε κάτω από το πρίσμα της σταθερότητας τιμών εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια για την οικονομία των κρατών μελών και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πολύ καλό λοιπόν το αποτέλεσμα. Ε, ε, το έχουν πετύχει η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία. Το καλύτερο που πέτυχαν εδώ και 15 χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι η εντολή μας, να επιτύχουμε τη σταθερότητα των ε, τιμών και αυτά είναι η πραγματικότητα που σας ανέφερα. Τώρα, για το μέλλον, οι παρατηρητές οι διάφοροι οικονομολόγοι, οι χρηματοοικονομικές αγορές προβλέπουν την ίδια ακριβώς σταθερότητα για το διάστημα των επόμενων 10 ετών. Αυτά είναι τα γεγονότα. Οι αριθμοί και οι προβλέψεις για το μέλλον. Αυτά τα είπα εν παρόδο. και όμως είναι πραγματικότητα. Και μένα με εκπλήσει αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα και θα συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το δρόμο. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων, αυτή είναι ένας διαφορετικός θεσμός. Εκεί δεν συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε και άλλα μέλη που προέρχονται από τις εποπτικές αρχές που σας ανέφερα και που προέρχονται επίσης από τον ακαδημαϊκό και τον επιστημονικό κόσμο προέρχονται από τις ε, εθνικές αρχές, είναι εθνικές εποπτικές αρχές. Αυτοί όλοι λοιπόν ενδιαφέρονται διακαώς να αξιολογήσουν τους ε, συστημικούς κινδύνους, να προβλέψουν ενδεχομένως κάποιες προκλήσεις που θα προκύψουν και αν και εφόσον χρειαστεί να καταθέσουν ε, συστάσεις για έγκαιρη προειδοποίηση. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι αυτός ο νέος θεσμός, ο νέος φορέας βρίσκεται πολύ κοντά στις ε, κεντρικές τράπεζες, στις εθνικές κεντρικές τράπεζες, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και νομίζω είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτό θα υπάρχει και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, γιατί ο συστημικός κινδυνός, επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αποφασίσατε τόσο εσείς εδώ όσο και το Κογκρέσο των Ηνωμένων αυτό το νέο φορέα να τον τοποθετήσετε κοντά στις κεντρικές τράπεζες διότι παίζονται μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμοι στόχοι. Οι φορείς αυτοί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και να επιδιώκουν την σταθερότητα. Αλλά να μην συγχαίουμε αυτά τα δύο πράγματα. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω και εγώ, έχετε πει κατά το παρελθόν ότι θα αναφέρεστε σε μας ε, ξεχωριστά και όχι στο πλαίσιο του νομισματικού διαλόγου. Και εγώ βέβαια πρέπει να επιβάλλω την πειθαρχία στα μέλη, να επιβάλλω τις σωστές ερωτήσεις, ε, ανάλογα με το με ποια ιδιότητα είστε εδώ, κάτι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Έπινγκ. Κύριε Τρισέ, κατά τη διάρκεια του τελευταίου ΕΚΟΦΗΝ, του Σεπτεμβρίου υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τον ε, φόρο χρηματοπιστωτικών, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η δική σας η άποψη ήταν απόλυτα σαφής. Υπήρξαν ε, άνθρωποι παρόντες ε, και είπατε ότι ο φόρος αυτός είναι πολύ κακή ιδέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θα αναγκάσει τις τράπεζες να μετακομίσουν αλλού από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Σανγκάη και το Χονγκ Κόνγκ. Ως εκ τούτου ε, θα πρέπει ο φόρος αυτός ε, να μην επιβληθεί. Συμφωνώ απόλυτα και παυξάνω κύριε Τρισέ. Ίσως λοιπόν μπορείτε για άλλη μια φορά να το επανεξηγήσετε το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή γιατί πάρα πολλά μέλη της Επιτροπής που βρίσκεστε είναι υπέρ αυτού του φόρου και ίσως μπορείτε να μας πείσετε με τη σοφία σας γιατί τελικά ο φόρος αυτός είναι τόσο κακή ιδέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε εγώ δεν τα είπα τόσο ωραία, τόσο ανάγλυφα όπως τα είπατε ότι δήθεν ε, θα μπορούσαν να υποφεληθούν οι αγορές. Αλλά είναι αλήθεια. Εγώ είπα, με βάση τις δικές μας αναλύσεις, πρόκειται για μία έννοια η οποία είναι απευκταία για οικονομικούς λόγους, για τεχνικούς γιατί θα υπάρξουν τεράστιες τεχνικές δυσκολίε στην επιβολή αυτού του φόρου και διότι αν τελικά εφαρμοστεί εδώ, κοιτάξτε, πρόκειται πάλι για την ίδια παρατήρηση που έχω κάνει για μια σειρά αλλαγών. Δηλαδή, οι αλλαγές πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμια κλίμακα. Και γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα, τουλάχιστον προς το παρόν. Γι' αυτό λοιπόν φοβάμαι ότι αν τελικά ο φόρος αυτός επιβληθεί εδώ, όποια και αν ήταν η πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση, απλά θα ανάγκαζε τις ε, οικονομικές συναλλαγές να λάβουν χώρα κάπου αλλού. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε μια συγκεκριμένη αγορά, αλλά θα μπορούσαν να μετατοπιστούν οπουδήποτε. Υπάρχουν τρεις λόγοι. Βεβαίως κατανοώ ότι είναι μια ιδέα η οποία μπορεί να είναι έτσι λίγο ελκυστική ιδιαίτερα ελκυστική και κατανοώ ότι Είναι αλήθεια ότι αρκετά κοινοβούλια, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι το ευρωπαϊκό, δεν θυμάμαι αν τοποθετηθήκατε από αυτού, αλλά πολλά εθνικά κοινοβούλια ε, ενστερνίζονται αυτό το φόρο τον επιθυμούν διακαώς, αλλά αυτό μας, μας δημιουργεί μας πολλές και μεγάλες δυσκολίες. Πράγματι, εγώ επιβεβαιώνω, δεν τα είπα όπως σας είπα τόσο πιστικά όπως τα αναφέρατε εσείς, αλλά εγώ πράγματι αναφέρθηκα ε, επιφυλακτικά για το θέμα αυτό στο ΕΚΟΦΗΝ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, ζητήσαμε από την Επιτροπή να αναφερθεί σε μία αξιολόγηση επιπτώσεων. Θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα τα υπέρ και τα κατά. Η επόμενη ερώτηση από τον Σφεν. Σφεν Γκίγκολντ. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε μια οικονομική συζήτηση για τα συν και τα πλήν του φόρου αυτού. Θεωρώ έτσι και αλλιώ ότι η φορολογική πολιτική είναι εκτός εντολής για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ω εκ τούτου δεν είναι και τμήμα της συζήτηση που πρέπει να γίνεται. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα έτσι ώστε το FTT αυτό να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Έχω μια άλλη ερώτηση όμως σχετικά με τα μαθήματα τα οποία παίρνουμε από την κατάσταση που σοβεί στην Ιρλανδία. Ανησυχούμε ιδιαίτερα. Οι διαφορές στα επιτόκια είναι, για τα ομόλογα ενώ είναι πάρα πολύ υψηλές. Αυτό δεν θα έπρεπε να ισχύει σε μια νομισματική ένωση. Ταυτόχρονα η Ιρλανδία ήταν πάντα ένα καλό παράδειγμα θα έλεγα, ένας καλός μαθητής σε σχέση με τις ρυθμίσεις αυτές. Τι έκανε η Ιρλανδία, μείωσε τις δημόσιες δαπάνες, μείωσε τους μισθούς, όπου μπορούσε το κράτος τουλάχιστον να το κάνει, το δημόσιο, και τώρα βλέπω ότι είναι η πρώτη χώρα η οποία έχει υποβαθμιστεί ε, με πάρα πολύ υψηλό ρυθμό. Λοιπόν, ε, ποιες είναι οι σκέψεις σας γύρω από αυτό, τι μαθήματα μπορούμε να βγάλουμε από την κατάσταση στην Ιρλανδία, τι συνέπειες θα έχει η κατάσταση στην Ιρλανδία γιατί και ποια είναι η δική σας προιπτική για να ξεφύγουμε από αυτήν τη δημοσιονομική κρίση. Η κατάσταση που υπάρχει στην Ιρλανδία τι συνέπειες θα προκαλέσει σε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης της αν συγκρίνει κανείς αυτά τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν από την Ιρλανδική κυβέρνηση στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, της μεταρρύθμισης φορολογικής πολιτικής και της μείωσης των δημοσίων δαπανών. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να πω, να επαναλάβω αυτό το οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ευρωζώνη και για τις μεμονωμένες χώρες. Πάντα λέμε ότι όταν βλέπουμε ότι βγαίνουμε από την ύφεση δεν φωνάζουμε νίκη. Αλλά ζητάμε να είμαστε επιφυλακτικοί για μια ακόμη φορά. Τώρα θα μπορούσαμε να πανηγυρίσουμε ότι ξεφύγαμε από την ύφεση, έτσι λένε οι δείκτες. έχουμε διορθώσει προς τα πάνω κατά 0,6% το ρυθμό ανάπτυξης για την Ευρωζώνη φέτος, αλλά παρόλα αυτά λέμε ότι αυτό δεν συνιστά νίκη και συστήνουμε επιφυλακτικότητα. Λοιπόν, αυτό το οποίο παρατηρήσαμε σε κάποιες χώρες είναι ότι ναι μεν έκαναν εξαιρετικές προσπάθειες όπως η Ιρλανδία η Ιρλανδία έχασε αναμονάδα σε ένα τεράστιο ποσοστό της ανταγωνιστικότητάς της τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια της περίοδου ανάπτυξης οικονομικής και μια ολόκληρη σειρά αποφάσεων που είχαν ληφθεί επέτρεψαν την ανάκτηση εν πολλής ε, της, ε, του κόστους αναμονάδας και την ανάκτηση κάποιων θέσεων στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Παρ' όλα αυτά η κρίση συνεχίζεται, η κατάσταση δεν είναι μια κατάσταση που ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στις 16, αύριο στις 17, είτε στις 27. Τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς και εμείς συστήνουμε σε όλες τις χώρες να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τις οποίες έχουν, γιατί οι δυσκολίες αυτές είναι διαφορετικές χώρα. Στην Ιρλανδία έχετε διαφορετικά προβλήματα από άλλες χώρες. Έχετε ένα τεράστιο χρηματοπιστωτικό τομέα και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι κάθε χώρα όπως και η Ιρλανδία έχει αποδείξει ιδιαίτερα η Ιρλανδία στο παρελθόν ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές και αυτό ακριβώς η κυβέρνηση της Ιρλανδίας και η Βουλή η Ιρλανδική κατανοούν ε, εξαίρετα στη φάση αυτή. Απευθύνουμε λοιπόν σε όλες τις χώρες να είναι επιφυλακτικές, να είναι πολύ προσεκτικές σχετικά με τις δικές τους οικονομικές πολιτικές, με, τις, ε, με τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζουμε, γιατί εξακολουθούμε να βιώνουμε μια κατάσταση η οποία είναι ιδιαιτέρως απαιτητική και απαιτεί να είμαστε όλοι ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλούτ. Δεν μπορούσα να σας βρω, σας έχασα εκεί πέρα που ήσασταν. Ευχαριστώ. Κύριε Τρισέ, ήθελα να ρωτήσω το εξή. Με πρόλαβαν κάποιοι συνάδελφοι. Ίσως όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, δεν ευχαριστήσαμε παρκώς την Ελλάδα που υιοθέτησε τόσο σκληρά ε, μέτρα ε, δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να θέσω μία ερώτηση. Είχα συμμετάσχει στην Γερμανία σε συζητήσεις με υπεύθυνου οικονομικών δήμων. Στην ε, Ρινανία Βεσφαλία, για παράδειγμα, ε, που είχαν υποστεί, είχαν δεχθεί τρομερές πιέσεις πέρσι. Φέτος η κατάσταση έγινε ακόμα δυσκολότερη και υπεύθυνη λένε ότι τα τρία τέταρτα των δημοσιονομικών προβλημάτων του σχετίζονται ακριβώς με την διεθνή χρηματοοικονομική κρίση και κατά συνέπεια δεν υπήρχε η δυνατότητα να προχωρήσουν παραπέρα λόγω των πιέσεων που υφίστανται ήδη. Το ερώτημα λοιπόν είναι μήπως υπάρχουν άλλες λύσεις, μήπως πρέπει να ακολουθούν άλλες λύσεις. Προφανώς αυτό κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερο ελκυστική για τους πολίτες. Πώς μπορεί, μήπως λοιπόν θα έπρεπε να βάλουμε στην ε, λύση της κρίσης της τράπεζας που ήταν ένα μεγάλο τμήμα των αιτιών. Τι να απαντάτε σε τέτοιους τοπικούς υπεύθυνου που δεν έχουν την ευθύνη της κρίσης αλλά την υφίστανται. Ευχαριστώ. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα ακριβώς τι είπατε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κάτι δεν κατάλαβα. Ποια είναι η συγκεκριμένη κριτική κατά της Ένωσης. Όχι, ε, δεν λέω, η ερώτηση που θέτουν οι πολίτες είναι γιατί εμείς στην κοινότητα, στο Δήμο, πρέπει σε τοπικό επίπεδο να πληρώνουμε μια κρίση για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται. Η πολιτική η οικονομική πολιτική που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δήμων. Να απαντήσω. Πρώτον, η κρίση είναι παγκόσμια. Δεν την δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση απεκάλυψε το, το, το, το εύθραυστο της παγκόσμιας οικονομίας. Παντού. Όχι ειδικά στην Ένωση. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση. Η παγκόσμια αυτή κρίση δημιουργεί προβλήματα. Και αυτό είναι ο λόγος τον οποίο εμείς ζητάμε από το χρηματοεπιστωτικό νέα να γίνει ανθεκτικότερος. Η κριτική, μεγάλο τμήμα της κριτικής κατά των νέων κανονιστικών, των νέων κανόνων που υιοθετήθηκαν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ήταν αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο, τελείω απαράδεκτο αυτή η κριτική, ακριβώς λόγω αυτών που είπατε. Ο κόσμος λέει σε εσά και σε όλες τις αρχές στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, δεν θέλουμε να ξαναδούμε την συνέχιση αυτής της ε, ευάλωτης και έφταυση κατάστασης του παγκοσμίου οικονομικού συστήματος που είδαμε μέχρι τώρα. Γι' αυτό η Ένωση και οι κυβερνήσεις, όχι μόνο της Ένωση, και η Αμερικανική κυβέρνηση και η Ιαπωνική κυβέρνηση έχουν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες ε, δυσκολίες. Είναι δυσκολίες για όλους μας. Εσείς είστε στην Ευρωζώνη, τουλάχιστον ένα θεσμικό όργανο έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει. Και το εξήγησε ότι είναι αξιοσημείωτο. Δεν περνάει ωστόσο στη δημοσιότητα τόσο δραστήριο όσο θα ήθελα. Αυτό είναι ένα στοιχείο ε, καθησυχασμού των πολιτών, των συμπολιτών μας. Η σταθερότητα των τιμών που τη θεωρούν πολύ σημαντική οι πολίτες. Δέχομαι απόλυτα ότι είναι πολύ δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες να είμαστε βέβαιοι ότι κάνουμε όλα όσα μπορούμε για να αποφύγουμε μια επανάληψη τέτοιας κρίσης. Είναι επίσης πολύ δύσκολο και το συζητούμε αυτό να είμαστε βέβαιοι ότι ε, όλες οι κυβερνήσεις θα κάνουν αυτό που απαιτείται για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα. Αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο. Ισχύει για την Ευρώπη. Το μήνυμα όμως τόσο και πάλι που έρχεται από την κατάσταση είναι το ίδιο για όλους. Και νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό να μετατρέψουμε σε αποδιοπομπαίο τράγο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όλοι ζούμε στην ίδια κατάσταση, όλοι βιώνουμε εξαιρετικέ συνθήκες, δεν είναι εύκολες, δεν διευκολύνει τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι τέτοιο, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών κυβερνήσεων, Το δέχομαι απόλυτα αυτό. Αλλά δεν πρέπει να μετατρέψουμε σε αποδιοπομπαίο τράγο κάποιο ευρωπαϊκό εθνικό όργανο, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο Σαραδράκος. Απευθυνόμενος στον κύριο Τρισέ, θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι εκτιμώ ιδιαίτερω τους χειρισμούς και τη συμβολή του στην επίλυση της κρίσης και στην αντιμετώπιση της κρίσης και ιδιαίτερα σε σχέση με το μνημόνιο για την Ελλάδα, τις ρυθμίσεις που έγιναν για την Ελλάδα. Είμαι Έλληνας Ευρωβουλευτής και τον ευχαριστώ. Θέλω να διαβεβαιώσω επίσης ότι στην Ελλάδα με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ελήφθησαν πάρα πολύ σκυρά μέτρα προκειμένου η χώρα να περιορίσει το τα δημοσιονομικά της ελλείμματα. Αλλά εκείνο το οποίο ε, κύριε Πρόεδρε, ε, με ανησυχεί είναι ότι πέρα από την ανάπτυξη την επιστημονική, την τέλεια επιστημονική ανάπτυξή σας, πρέπει να δούμε και το θέμα πολιτικά. Διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλη η Ευρώπη και κυρίως οι λαοί της Ευρώπης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Είδατε τι έγινε προχθές στη Γαλλία, βλέπουμε συνεχείς απεργίες και προβλήματα και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα του Νότου. Πέραν όμως από την δημοσιονομική πειθαρχία και τις κλασικές μεθόδους για μια ταχύρυθμη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα κτλ. Εκείνο το οποίο με φοβίζει κύριε Πρόεδρε είναι ότι σημαντικό στοιχείο της κρίσης είναι οι λεγόμενες αγορές οι οποίες φαίνεται ότι δεν αυτορυθμίζονται. Και δεν είναι το θέμα νομικό ή ποινικό. Πρέπει να αντιμετωπιστούν με οικονομικές κινήσεις κατά την άποψή μου. Και θα σας παρακαλούσα στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται για τη νέα ρυθμιστική αρχή να λάβετε μέτρα εις τρόπον ώστε να εξισορροπήσει η επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος με την κοινωνική αντιμετώπιση του θέματος. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις αγορές δεν νομίζω ότι ό,τι άλλο και αν καλύψουμε θα έχουμε ελληματικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I, of course, uh, Συμφωνώ αναμφισβήτητα με όλα αυτά που είπατε, αλλά θα ήθελα να επιτρέψετε να πάω λίγο πιο πέρα, να επεκτείνω αυτά που είπατε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα όπου αυτή η ισορροπία ανάμεσα σε ελευθερία και ρυθμίσεις. Ε, ρύθμιση τραπεζών, ε, μη τραπεζών, συνταξιωτικών ταμείων, ασφαλιστικών φορέων και πολλών άλλων. Όλα αυτά τώρα πλέον συζητούνται όχι μόνο μέσα στην Ευρώπη, όχι μόνο στον εκβιομηχανισμένο κόσμο, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο και με τις αναδυόμενες χώρες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να εκπονήσουμε τις κατάλληλες ε, προδιαγραφές και τις ρυθμίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, τότε θα προκαλέσουμε περαιτέρω αστάθεια θα έλεγα μάλιστα ίσως και ακόμα μία κρίση και ίσως και μετατόπιση των δραστηριοτήτων, κάτι που δεν μας συμφέρει που δεν είναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πράγματι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση η οποία απαιτεί ιδιαίτερη σοφία ε, εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα. Και εγώ ο ίδιος το βιώνω αυτό, το βλέπω βλέπω αυτές τις ε, ασύλληπτες αλλαγές που υπάρχουν στην ε, διασύνδεση των οικονομιών του κόσμου και από τότε που εμφανίστηκε η κρίση και ο αναδιόμενος κόσμος πλέον συμμετέχει σε όλη αυτή τη συζήτηση. Στην ομάδα των G20 έχουμε έτσι μια συμβολική ε, παράσταση αυτής της κατάστασης, αλλά θα έλεγα παρόλα αυτά ότι έχουμε έτσι μια ε, σιωπηρή επανάσταση σε όλες τις συζητήσεις ε, που λαμβάνουν χώρα. Και υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο είμαι σίγουρος και ο κύριος Αλαβράκος φαντάζομαι θα συμφωνήσει μαζί μου. Οι λαοί μας δεν θα μας συγχωρήσουν αν για δεύτερη φορά βιώσουμε την ίδια τραγωδία. Δεν θα μας ε, συγχωρήσουν ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στην Ευρώπη, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη προηγμένη κοινωνία ή οικονομία. Άρα δηλαδή είμαστε καταδικασμένοι να βρούμε ε, τις λύσεις εκείνες που θα καταστήσουν το σύστημα περισσότερο ανθεκτικό, τούτο όμως προϋποθέτει προσπάθειες και μερικοί βέβαια δεν είναι ευχαριστημένοι με τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν. Ο κύριος Μάρτιν, Hans Peter Martin. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να διαβάσω μία παράθεση και διαβάζω το καθοριστικό σημείο παραμένει πως ε, ένας ε, κόσμος ε, μπορεί να εμφανίζεται χωρίς έντονη μόχλευση. Πώς είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη. Deleveraging σε τελική ανάλυση σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να περιοριστούν σε ένα τέτοιο επίπεδο χρέους ε, το οποίο να μπορούν να εξυπηρετήσουν και σε περιόδους κρίσης. Εάν η ανάπτυξη περιοριστεί αναγκαστικά μειώνονται και τα περιθώρια. Αυτή είναι η παράθεση και ερωτώ κύριε Πρόεδρε, εσείς συμφωνείτε με αυτό, συμφωνείτε με αυτήν την εικόνα που θα έχουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Ευρωζώνη με όλες τις συνέπειες. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω αυτή η διαδικασία του deliveraging της απομόχλευσης ε, που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει μόνο στην Ευρωζώνη, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις Ηνωμένε Πολιτείες... και σε άλλα μέρη του κόσμου. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία η οποία κατόρθωσε να αυξήσει τη μόχλεψη και έτσι φτάσαμε στην κρίση που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα δηλαδή αυτό που ίσως πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν από αυτού. Αυτό λοιπόν που οφείλουμε να κάνουμε είναι στην παγκόσμια οικονομία να εντάξουμε και αντικυκλικά στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν να αποφύγουμε αυτή την υπερβολική μόχλεψη η οποία πάντα συνοδεύεται από υπερβολική απομόχλευση. Έχουμε λοιπόν ε, αυτές τις ε, εκρήξεις ε, που πολύ συχνά χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της οικονομίας, αλλά αυτό που βιώνουμε τώρα είναι η χειρότερη πτώση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατ' ουσίαν δηλαδή αντιμετωπίζουμε κάτι, ένα ακραίο φαινόμενο και προέκυψε αυτό μετά από μία περίοδο έντονης μόχλευσης που ήταν και αυτή η πιο έντονη, η, πιο, η ακραία, πλέον ακραία που υπήρξε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα δηλαδή πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επιδιώξουμε μια τέτοια εξέλιξη, εθνική και παγκόσμια, που δεν θα είναι τρωτή σε πιέσεις. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να απαντήσει κανείς σε αυτό. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι ως το δυνατόν περισσότερο να αποφύγουμε προκυκλικούς μηχανισμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται μέσα στα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά. Έχουμε κεφαλουχικές απαιτήσει, οι οποίες από μόνες τους μπορεί να είναι αντικυκλικές. Και Αυτό το ανέφερα ως ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πάντως όλα αυτά δεν είναι εύκολα, αλλά είναι όμως απαραίτητα. Ο κύριος Φέιο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε Τρισέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω να σας ευχαριστήσω για τον σαφή τρόπο με τον οποίο ε, αντιμετωπίσετε το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης και να σας πω ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει απόλυτα την μια ευρωπαϊκή, σαφή και αποτελεσματική λύση με συγκεκριμένους σαφείς και σημαντικούς ρόλους για την τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Εταιρική Τράπεζα και το Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θέλω να ρωτήσω, Πρόεδρε, μέχρι πού πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει η αξιολόγηση της Επιτροπής των ε, προϋπολογισμών των κρατών. Μιλήσαν, έγινε λόγος για ανάλυση των μεγάλων στοιχείων, τα, των γενικών στοιχείων δηλαδή. Ποια είναι αυτά τα γενικά στοιχεία. Είπατε επίσης ότι πρέπει να έχει συστάσεις προς τα κράτη σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα. Σας υπενθυμίζω την Πορτογαλία. Τα, οι δημόσιες δαπάνες αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα ελέγξιμες. Χρειαζόμαστε να πληρώσουμε πολύ μεγάλα επιτόκια. Τι ανταγωνιστικότητα, τι συστάσεις ανταγωνιστικότητας μπορείτε να δώσετε σε ένα κράτος που αντιμετωπίζει τέτοια κατάσταση κύριε Τρισέ. Πρώτα-πρώτα, το ενδιαφέρον του, της έννοιας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι ότι βλέπεις τις δυσκολίες όσο πιο νωρίς γίνεται και συνδέεις τα άλλα κράτη στην εξέταση μιας κατάστασης συνολικά με τρόπο ευθύ, ειλικρινή όλες οι χώρες μέλη της Ένωσης ξέρουν ότι είναι ότι μία εξαρτάται από την άλλη, ότι είναι αλεξαρτώμενες. Ως τμήματα της ενιαίας αγοράς. Οι δε χώρες της Ευρωζώνης ξέρουν ότι εξαρτώνται ακόμη περισσότερο η μία από την άλλη λόγω και της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου νομίσματος. Και το είδαν. Τι σημαίνει κάτι τέτοιο με την πίεση της κρίσης. Άρα υπάρχει βούληση και περιμένω να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό εξάμεινο όσο καλά γίνεται. Δεν θα μπω τώρα στην θέση της Επιτροπής. Είναι σαφές ωστόσο ότι όπως είπα από το 2005 συστήσει εντονότατα στα μέλη της ζώνης ευρώ να εφαρμόζουν αυστηρά το σύμφωνο, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Δυστυχώς δεν το έκαναν. Παρότι το ζητούσαμε και εμείς και η Κομισιόν. Και κάποιες χώρες και το Κοινοβούλιο το ζητούσαν. Ζητάμε επίσης όμως να υπάρχουν, να τηρούνται και οι δείκτες ανταγωνιστικότητας απόλυτα. Οι εσωτερικές και εγχώριες ανισότητες μόνο έτσι μπορούν να καλυφθούν, διότι θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό σε έναν χώρο ενιαίου νομίσματος το, το ορόσημο είναι ξεκάθαρο. Το μήνυμα που περνάμε είναι 11,5 χρόνια λιγότερο από 2%. Τα επόμενα φέτος κοντά στο 2%. Τα επόμενα 11 χρόνια κάτω ή κοντά από το 2%. Ξέρετε που βρίσκεστε. Άρα οι αποφάσεις σας πρέπει να στηρίζονται στο γεγονός ότι είστε τμήμα αυτής της τεράστιας υπήρου σταθερότητα. Αν τώρα ο εθνικός πληθωρισμός είναι υψηλότερος από το μέσο όρο, αν οι ονομαστικές εξελίξεις προχωρούν γρήγορα, τότε μειώνεται η ανταγωνιστικότητα και δημιουργούνται προβλήματα μετά από ένα χι χρόνο. Αυτό είναι το μήνυμα για όλες τις χώρες, την Πορτογαλία και όλες τις άλλες. Η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε, μια και ήλθε η συζήτηση και στην Ελλάδα, θα ρωτήσω και εγώ κάτι που έχει σχέση με τη χώρα μου. Ήθελα να σας πω καταρχάς πώς κρίνεται μετά από τα σκληρά μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας που έχουν εφαρμοστεί την υστέρηση των εσόδων. Είναι περιττό να αναφερθώ το πόσο μας ανησυχεί αυτό για τις οικονομικές, κοινωνικές συνέπειες αλλά και την επίτευξη των στόχων της δημοσιονομικής εξυγίανσης, η υστέρηση των εισόδων των εσόδων. Και το δεύτερο ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι τα δημοσιεύματα στον ελληνικό και στον διεθνή τύπο για την ε, ε, ε, επέκταση μη του μνημονίου μετά το 2013. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντίθετη προς αυτό το ενδεχόμενο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δείχνει πρόθυμο. Ήθελα να ξέρω εσείς, σαν τρίτος δανειστής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ποια είναι η άποψή της και αν πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση έναντι των, ε, της ε, κοινή θέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διεθνώς Νομισματικό Ταμείου, διότι η ασάφεια αυτή δεν ωφελεί ούτε τις εθνικές προσπάθειες, ούτε τους στόχους που πρέπει να πιάσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να διευκρινίσω για μια ακόμη φορά. Θα ζητούσατε από τον Μπερνάνκε σαν παράδειγμα να σας πει αν για το Τέξας, τη Μασαχουσέτη, την Αλάσκα ή την Καλιφόρνια κάποια πολιτεία κάνει κάτι καλό ή δεν κάνει αυτό που πρέπει. Κοιτάξτε, εμεί είμαστε πάνω κάτω στη θέση του Federal Reserve. Εμείς ζητάμε από κάθε μέλος να παίρνει τι αποφάσεις 16 χώρες σήμερα, 17 αύριο, 330 περίπου εκατομμύρια από την 1η Ιανουαρίου του 2011. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζάς μας είναι εμπειρογνώμων για όλους. 330 εκατομμύρια. Έχει το ίδιο δικαίωμα ψήφου. Μία ψήφος, ένα μέλος. Είτε είναι από την Κεντρική Τράπεζα της τάδε χώρας ή της δίνα χώρας, ανεξάρτητα από τις διαφορές τις πληθυσμιακές. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορές πληθυσμιακές ανάμεσα σε χώρες, ένα προς 50, ένα προς 100 κτλ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Mm. Και υπάρχει βέβαια και το διευθυντικό κομμάτι. Το Διευθυντικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών σε μία ήπειρο 330 εκατομμυρίων πολιτών. Σε ένα σύνολο 330 εκατομμυρίων πολιτών. Έχετε τις κυβερνήσεις απ' την άλλη, οι οποίες είναι υπεύθυνε για τις δικές τους πολιτικές. Έχετε το Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία αυτών των πολιτικών. Σύμφωνα με τη συνθήκη δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα επιβλέπουν το τι κάνουν οι κυβερνήσεις. Υπάρχει το Συμβούλιο, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αξιολογεί τις καταστάσεις και κάνει τις απαιτούμενες προτάσεις. Και εμεί λοιπόν απευθύνουμε έκκληση σε όλα αυτά τα θεσμικά όργανα να έχουν ένα κοινό προσανατολισμό και να συνειδητοποιήσουν το ύψος των ευθυνών τις οποίες πρέπει να αναλάβουμε. Δεν είναι άχρηστο να το υπενθυμίζω αυτό γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε. Βέβαια κάτω από ειδικέ συνθήκες και εμείς εκφραζόμεθα και εμείς δίνουμε τις δικές μας συστάσεις αν θέλετε. Αλλά παρόλα αυτά η ευθύνη μας είναι σε επίπεδο υπηρετικό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερωτήσεις τις οποίες πολλές που μου κάνετε θα πρέπει να τις κάνετε τις ερωτήσεις αυτές είτε στο Συμβούλιο, είτε στην Επιτροπή, είτε στις επιμέρους κυβερνήσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να πω πάντως είναι ότι έχουν υπάρξει σημαντικότατες αλλαγές στην τροχιά της ε, ε, πολιτικής της συγκεκριμένης χώρας, της Ελλάδας. Έχουν ζητήσει, εμείς έχουμε ζητήσει να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές. Υπήρξαν τέτοιες οι αλλαγές, εμείς θα αξιολογήσουμε αν θέλετε τους προσανατολισμούς αυτούς και τη σοφία τους σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το μήνυμά μου τώρα σε αυτή τη φάση, το μοναδικό μου μήνυμα είναι εφαρμόστε αυστηρά αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί, τα οποία είναι σωστά προσανατολισμένα και τα οποία αξιολογούνται ανατρίμηνο όπως γνωρίζετε και από το ΔΝΤ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εάν αυτό γίνεται καλά, όπως πιστεύουμε ότι θα γίνει καλά, αν αυτό γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο, τότε περιμένω ότι αυτό θα γίνει αντικείμενο αναγνώρισης και θα αλλάξει μια κατάσταση αξιολόγησης η οποία προοδευτικά σταδιακά έχει αρχίσει να αλλάζει. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Χακμάρκ. Τα συστήματά μας πρέπει να είναι ανθεκτικά, όπως είπατε. Για να υπάρξουν όμως ανθεκτικά δημοσιονομικά συστήματα, πρέπει να έχουμε σταθερές, ε, σταθερά οικονομικά μεγέθη σε επίπεδο δημοσιονομικό και ισχυρές οικονομίες κρατών μελών. Μπας Σήμερα έχουμε ας πούμε ένα μέσο όρο ελλημάτων, 7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσο όρο λέμε. Και μπορεί να έχουμε και μία μείωση κατ' έτος 1%. That is the 2020 and uh, a decade of austerity. But at the same time we need... Ταυτόχρονα όμως η μείωση των ελλημάτων δεν αρκεί, απαιτείται και ανάπτυξη. Και αυτό ε, απαιτεί αν θέλετε και άλλους ε, τομείς παρέμβασης και άλλες μεταρρυθμίσεις γιατί το θέμα των πολιτικών λιτότητας, των αυστηρών πολιτικών λιτότητας βλέπουμε ότι παρουσιάζουν κινδύνους, δημιουργούνται προβλήματα πολλές φορές από τις πολιτικές αυτές. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσετε να μας δώσετε κάποιες σκέψεις για το αν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις χρηματαγορές με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, μια δεύτερη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση η οποία θα συνοδεύεται και από ε, πολιτικές ε, αυστηρές λιτότητας. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία η οποία μερικές φορές να είναι αντιφατική σε σχέση με τα μέτρα που παίρνουμε, με τα αριθμιστικά εννοώ μέτρα. Σας ευχαριστώ κύριε Χεκμάρκ. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω, λέει ο κ. Τρισέ. Πρώτη, για τις οικονομικές πολιτικές. Ή μιλήσατε για κάποια τάξεις μεγέθους των ελλημάτων. Θυμίστε, ενθυμίστε ίσως όταν συζητούσαμε για τη συνθήκη του Μάστριχτ είχαμε πει το 3% ένα όριο το οποίο πολλοί είχαν θεωρήσει υψηλότατο. Βλέπουμε όμως ότι ο μέσος όρος τώρα πλέον είναι πολύ υψηλότερος. Προφανώς όλα αυτά εξηγούνται. Εξηγούνται γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε όπως είπα και προηγουμένως τη χειρότερη οικονομική κρίση από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το να πιστεύει όμως κανείς ότι όταν είναι σε επίπεδο μέσου όρου 7% ή και υψηλότερον του 7% βρίσκεται στην ίδια κατάσταση σαν να ήταν σε μείον 2 αντί για 7% δεν έχει λογική. Σε αυτή την περίπτωση αν δεν κάνεις τίποτα χάνεις την εμπιστοσύνη στις αγορές, τα νοικοκυριά δεν καταναλώνουν, φοβούνται, γνωρίζουν ότι θα έχουν σοβαρά προβλήματα και με τη φορολογία, οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν και οι επενδυτές και αποταμιευτές και αυτοί δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στο τίμημα το οποίο καλούνται να πληρώσουν. Συνεπώς λοιπόν, το πραγματικό αντίμετρο δεν θα είναι να πούμε ότι αν δεν κάνουμε τίποτα ή αν ακόμα και αυξήσουμε λίγο το έλλειμμα τότε θα βρεθούμε σε καλύτερη φάση. Αυτά είναι τα λεγόμενα γραμμικά μοντέλα. Νομίζω ότι το αντίμετρο θα είναι ότι αν δεν κάνουμε τίποτα τα πράγματα δεν μπορεί παρά να χειροτερεύσουν. Πρέπει να το χωνέψουμε αυτό. Είναι σαφές αυτό. Βέβαια δέχομαι ότι στο παρελθόν είχαμε αγνοήσει την αντίθετη λογική. Εγώ δεν λέω ότι τώρα πια αγνοείται η λογική αυτή στην οποία αναφερθήκατε. Υπάρχει γενική αναγνώριση και σε επίπεδο 27 ότι το θέμα της εμπιστοσύνης στην οικονομία στο μέλλον είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε και να καλλιεργήσουμε. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα στο οποίο και εσείς αναφερθήκατε, είναι το θέμα της ρύθμισης. Εφόσον ενισχύσουμε, καταστήσουμε πιο αυστηρά τα στάνταρτς και τις ρυθμιστικές αυτές αποφάσεις, αυτό κάνουμε το τελευταίο καιρό και συνεχίζουμε να κάνουμε, μήπως εμποδίσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας. Αν διαβάσετε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα πιο γνωστά, θα δείτε εδώ να αντικατοπτρίζονται και οι δύο ανησυχίες. Κάποιοι μας λένε ότι είσαστε πάρα πολύ δειλοί, είσαστε πολύ ντροπαλοί σε εισαγωγικά. Και δεν θα γυρίσουμε στο 2008 ξανά, δεν θα έχουμε ένα σύστημα τόσο εύθραστο. Κάποιοι πιστεύουν λοιπόν ότι θα πρέπει να σκληρύνουμε ακόμα περισσότερο το, τις, τους ορισμούς που χρησιμοποιούμε για το κεφάλαιο και τις ε, κεφαλαιοκές απαιτήσεις κτλ. Από την άλλη, κάποιοι λένε ότι υπερβάλλουμε στις ρυθμίσεις και ότι θα παρεμποδίσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας. Γιατί δεν θα είναι δυνατόν να υπάρξει η νέα αυτή χρηματοδότηση, θα δημιουργήσετε μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση λόγω ακριβώς της σκληρότητας των νέων ρυθμίσεων τις οποίες επιβάλλεται. Και αυτό το οποίο εμείς τελικά προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στις δύο λογικές. Να είμαστε έλογα και εύλογα θα έλεγα βέβαιοι για τα μέτρα μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια ενός σταθερού καθεστώτος θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, να καταστήσουμε ισχυρότερο το σύστημα και να μπορέσουμε επίσης να διαβεβαιώσουμε το κοινό ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ότι το πιστοτικό ε, σύστημα ε, δεν κινδυνεύει όπως πίστεψαν κάποιοι ότι κινδυνεύει και υπάρχει μια μεταβατική περίοδος τα πλαίσια της οποίας πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουμε τις τάσεις για την ανάκαμψη. Λοιπόν, αυτή είναι η προσπάθεια εξισορρόπησης των πολιτικών μας. Ε, συγγνώμη, αλλά ήταν η ερώτηση πάρα πολύ σε εισαγωγικά τολμηρή. Περνάει η ώρα. Ε, πρέπει να έχουμε κατά νου και τους άλλους που θα ακολουθήσουν και θα υποβάλουν ερωτήσεις. Ο Λεωνάρντο. Πρόεδρε, στην ε, σημερινή σας ε, παρουσίαση, κυρίως όσον αφορά τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις, εσείς προβήκατε σε θετική αξιολόγηση, αν κατάλαβα καλά, τουλάχιστον για τις εξελίξεις κατά το δεύτερο τρίμηνο. Και σε αυτή σας την αξιολόγηση οι εξαγωγέ και η εσωτερική ζήτηση ε, στην Ευρωζώνη πόσο έπαιξε ρόλο. Στο δεύτερο σκέλος ε, τη σκέψη σα για τι οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις, εκεί όμως εσείς ήσασταν ιδιαίτερα επιφυλακτικό. μιλήσατε για επιβράδυνση ρυθμού, ε, για ασάφεια. Για ποιο λόγο το πράξατε αυτό. Ίσως για τις εξελίξεις του ευρώ και τις εξαγωγές, επιπτώσεις εξαγωγές. Εν πάση περιπτώσει, οι αλλαγές, αν δεν είναι ισορροπημένες, μήπως πιστεύετε και εσείς ότι θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική ζήτηση και στις, ε, στις κοινωνικές ανάγκες γενικότερα, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει άμεση σχέση με την επαναφορά της εμπιστοσύνη κάτι το οποίο εσείς αναφέρετε πολύ συχνά. Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, Κατά το δεύτερο τρίμηνο διαπιστώσαμε ότι υπήρξε μεγαλύτερη επιβράδυνση ανάπτυξης από ό,τι αναμένετο. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εσωτερική ζήτηση και πολύ λιγότερο στην εξωτερική ζήτηση. Για το 1% Το 0,1% οφείλεται στην εξωτερική ζήτηση. Υπήρξε δηλαδή ε, κάποια θετική συνεισφορά, αλλά αρκετά περιορισμένη. Είχαμε λοιπόν 0,1% συνεισφορά από την ε, εξωτερική ζήτηση, το 0,2% από τα αποθέματα και το υπόλοιπο από την εσωτερική ζήτηση δηλαδή επενδύσεις ε, και ιδιωτική κατανάλωση. Αυτή ήταν η κατάσταση. Θα δούμε τώρα τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν μπορώ όμως ε, να ισχυριστώ ότι όλα αυτά ε, προέκυψαν γιατί είχαμε πάρα πολύ καλές εξελίξεις στο εξωτερικό σκέλος, ότι γι' αυτό ε, βιώσαμε ανάπτυξη. Τώρα βέβαια είμαστε πολύ προσεκτικοί για τις αναλύσεις που κάνουμε. Εκεί δεν βλέπουμε να προκύπτουν ε, ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά το προφίλ της μελλοντικής ανάπτυξης. Και επιτρέψτε μας να αναφέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αναθεωρήσαμε προς τα άνω την ανάπτυξη για την εφετινή χρονιά και από περίπου ένα για εφέτος καταλήγουμε στο περίπου 1,6. Άρα δηλαδή μια αλλαγή προς τα πάνω που είναι σημαντική. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το προφίλ της ανάπτυξης για του χρόνου ότι έχει δίθεν αλλάξει αυτό. Για την επόμενη χρονιά θα μιλάμε πάλι για την ίδια τάξη μεγέθους, παίρνω πάντα το μέσο όρο, από 1,2 στο 1,4 και αυτό το συν 0,2% προέρχεται εκ μεταφοράς από το 2011 10 στο 2011. Διότι, όπως σας είπα, αναθεωρήσαμε προς τα πάνω τη μέση ανάπτυξη κατά το 2010. Βλέπετε λοιπόν, ε, πρέπει να παραμείνουμε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και συνετοί. Πράγματι, ε, διαπιστώσαμε ότι είχαμε υποτιμήσει την ανάκαμψη, όμως πιστεύουμε ότι δεν θα ήταν σωστό να ε, βγούμε διθυραμβικά και να πούμε ότι να τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου βιώνουμε ουσιαστική ανάπτυξη. Όχι, πρέπει να παραμείνουμε επιφυλακτικοί. Νομίζω ότι αναφέρθηκα ε, στο θέμα των μελλοντικών τριμήνων και για μένα τουλάχιστον Ορμόμενος από την ερώτηση θα ήθελα να πω ότι πρέπει να αυξήσουμε το δυναμικό μας της ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε ουσιαστική δημογραφική ανάπτυξη. Και αυτό είναι θέμα κλειδί. Αν πάρουμε την ανάπτυξη κατά κεφαλή στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Ευρωζώνη ή στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, που δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά πάρουμε την Ευρωζώνη. Μιλάμε 1% αύξηση κατά κεφαλή τα τελευταία 10 χρόνια στην ε, Ευρωζώνη και 1,1% στις Ηνωμένε Πολιτείες. Επειδή όμως οι Ηνωμένε Πολιτείες η δημογραφική ανάπτυξη είναι πολύ δυναμικότερη, τα στοιχεία κατ' ουσίαν είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη στις Ηνωμένε Πολιτείες από ό,τι στην Ευρώπη και τούτο λόγω δημογραφίας. Εδώ πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα της ε, ανάπτυξης, της ε, αύξησης της ανάπτυξης και για μας η λύση είναι συνεχείς διαρθρωτικές αλλαγές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, εγώ χαίρο διότι η τράπεζα ξεκίνησε non-standard measures, άτυπα, έκτακτα μέτρα που είναι συμβατά με, τις, με τους στόχους της τράπεζας και βελτιώνουν την ε, λειτουργία της ε, τράπεζας ε, σε τομείς που δεν λειτουργούσαν καλά. Υπάρχει βέβαια μια σειρά κινδύνων. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να υλοποιηθούν. Δεύτερο ερώτημα. Η μεταρρύθμιση, η γενική μεταρρύθμιση ενώπιον της κρίσης. Δεν θεωρώ ότι εσείς είσαστε κάθετα αντίθετο με ένα φόρο φόρο χρήματο-οικονομικών συναλλαγών, αλλά έχετε κάπω έτσι ε, μια θέση με περισσότερες αποχρώσεις. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι φόροι που θα συνοδεύονται από, από ε, έλεγχο και δημοσιονομική παρακολούθηση. Μήπως μαζί με τον έλεγχο και την εποπτεία θα μπορούσαμε να δούμε και τις δυνατότητες αυτής της ε, εφαρμογής ενός φόρο που θα αποτελούσε μια πληρέστερη απάντηση στην κρίση. Thank you very Ευχαριστώ. Σε αυτά τα μη τυπικά μέτρα, τα non-standard measures, νομίζω ότι είναι σχεδιασμένα για να επιτρέπουν σε εξαιρετικές καταστάσεις οι μηχανισμοί διαβίβασης νομισματικής πολιτικής να λειτουργούν όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε αυτά τα εξαιρετικά μέτρα που είναι η άνευ περιορισμού παροχή ρευστότητας σε σταθερό επιτόκιο που γενικεύσαμε μετά την εντατικοποίηση της κρίσης κατά, μέσο του, κατά μέσα του Σεπτεμβρίου του 8 και τα άλλα μέτρα μεταξύ των οποίων και την, την, ε, τις αγορές ακάλυπτων ομολόγων και τις αγορές ε, ομολόγων από την τράπεζα. Ό,τι κάνουμε λοιπόν σχεδιάστηκε για να επιτρέπει τη σωστή μεταφορά, μεταβίβαση οδηγιών οριζοντικής πολιτικής. Πιστεύουμε ότι τα τυπικά μέτρα, τα standard measures, πάντα πρέπει να είναι αντίστοιχα στον βασικό μας πρωταρχικό στόχο, τη σταθερότητα των τιμών. Να είναι αξιόπιστε σε αυτό το στόχο, αυτή είναι η εντολή μα, αυτό ζητά από εμά ο λαό τη Ευρώπη και αυτό είναι που είναι καλό για τη συνολική χρηματοοικονομική σταθερότητα. Γιατί αν δεν είχαμε τις προσδοκίες σταθερότητας τιμών και την σταθερότητα των τιμών θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη φορολογία σε συναλλαγές, σε τράπεζες κλπ. Επαναλαμβάνω ότι δεν υποστηρίζουμε την φορολόγηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Για τις τράπεζες πάντα λέγαμε ότι πρέπει πρώτα να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν νέα standards και επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση που θα ήταν τα ενδεδειγμένα και τα αντίστοιχα ώστε να επιτρέπουν στον κλάδο να είναι πολύ λιγότερο τρωτός και πολύ πιο ανθεκτικός, άπαξ και γίνει κάτι τέτοιο, οι κυβερνήσεις, ορισμένες ή διάφορες κυβερνήσεις μπορεί να αποφασίσουν, να θέλουν, να ξεκινήσουν φορολογία οι, τρα, οι χώρες είναι σε διαφορετικές ε, καταστάσεις, υπάρχουν διαφορετικές θέσεις και στην Ευρώπη και εκτός. Καταλαβαίνω ότι κάθε θέση στην ουσία καθοδηγείται από την πρόσφατη εμπειρία. Όταν η πρόσφατη εμπειρία ήταν ιδιαίτερα δραματική και έπρεπε να, χρηματο να χρηματοδοτήσει ο φορολογούμενος στις τράπεζες το αίτημα για φορολόγηση των τραπεζών είναι ισχυρό, εκεί όπου δεν υπήρχαν τέτοιες εμπειρίες, το αίτημα είναι πολύ λιγότερο ισχυρό. Ευχαριστώ. Uh, δεν έχουμε πλέον καθόλου χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, υπογραμμίσατε στις uh, εισαγωγικές σας παρατηρήσεις την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στις uh, Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρώπη. Η συνάντηση των 20 μας έδωσε την αίσθηση ότι αυτό όλοι το επιθυμούν. Λέει ο κ. Κλίντς, να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα πλαίσια μιας κρίσης η οποία είναι σφαιρική. Μετά από δύο χρόνια, βλέποντας το τι έχει γίνει στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρώπη, υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Υπάρχουν ελάχιστες ομοιότητες, αλλά και πάρα πολλές διαφορές. Απογοητεύομαι για αυτές τις διαφορές. Δεν μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για άποψη της ομάδας των 20 εδώ. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στη χώρα μου, στη Γερμανία, τράπεζες οι οποίες σώθηκαν από την κυβέρνηση, ανήκουν στην κυβέρνηση και πληρώνουν εκατομμύρια μπόνους στα στελέχη τους. Ενώ είχαν πεθάνει σε εισαγωγικά εδώ και λίγο καιρό. Λοιπόν, έτσι οι πολίτες ε, βλέπουν ότι κανένας δεν πήρε το μαθημά του και ότι τα πράγματα παραμένουν τα ίδια. Δεύτερον, ε, αυτές οι ρυθμίσεις οι οικονομικές, το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό, χρηματοπιστωτικό μέσο μάλλον, σε τρία χρόνια θα έχει λήξει ουσιαστικά. Λοιπόν, κανένας δεν έχει συμφέρον η Ελλάδα, η Ιρλανδία να αντιμετωπίσουν ε, τα ίδια προβλήματα εκ νέου με αυτά που αντιμετώπισαν πριν μερικούς μήνες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν το μέσο αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί ή αν θα πρέπει να υπάρξει ένας νέος μηχανισμός αναδιάρθρωσης ο οποίος θα πρέπει να συζητηθεί. Για το πρώτο θέμα. Θα συμφωνήσω μαζί σας λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πλαίσια των δημοκρατιών μας να είμαστε βέβαιοι ότι όλα όσα γίνονται και όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται είναι μέτρα τα οποία συναντούν μια διεθνή παγκόσμια συνένεση. Ίσως είναι λίγο δύσκολο αυτό. Είστε λίγο αυστηρός. Διαφορές ανάμεσα σε εμά και στην Αμερική υπάρχουν. Ας δούμε κάποια παραδείγματα. Η Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου. Δεν τέθηκε το θέμα αυτό στα πλαίσια της λογικής που λέει ότι θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά λεπτομερώς με τις Ηνωμένε Πολιτείε. γιατί έχουμε τον ίδιο το δικό μας πολιτισμό, έχουμε ένα ίδιο πολιτισμό, ίδιες παραδόσεις θα έλεγα. Φυσικά πολλά πράγματα είναι τα ίδια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και υπάρχουν ε, εμπνεύσει θα έλεγα οι οποίες ε, είναι κοινέ και στις δύο πλευρές. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν κάποιες ρυθμίσεις επιμέρους οι οποίες ήταν πιο ξεχωριστές και πιο χαρακτηριστικές για τη μία πλευρά ή την άλλη όπως η Επιτροπή αυτή να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να είσαστε λίγο πιο, θα έλεγα, λιγότερο απόλυτο σε σχέση με τον συντονισμό αυτά τα οποία συζητιούνται για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία των πιστοτικών ιδρυμάτων δεν συζητιούνται μόνο με τις Πολιτείες αλλά και με τις ανερχόμενες χώρες. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα, τα πράγματα δεν είναι πολύ απλά, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα αρνητικοί. Η προσπάθεια που γίνεται είναι περίπλοκη, είναι προσπάθεια που δεν αποδίδει αμέσω και πρέπει να συνεχιστεί. Για το μέσο αυτό, Κανονικά ε, θα πρέπει εμείς μέχρι τη χρήση του συγκεκριμένου μέσου να αλλάξουμε τα πράγματα τώρα, σήμερα να αλλάξουμε τα πράγματα και στις ε, μακροπρόθεσμες πολιτικές μας και στις άμεσες οικονομικές πολιτικές σημασία έχει να αλλάξουν τα πράγματα τώρα. Να πούμε ότι εμείς ε, έχουμε ένα σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε και αυτό βέβαια στην περίπτωση κατά την οποία δυστυχώς υπάρξουν τέτοιου είδους κρίσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, καθυστέρησα να έρθω. Παρακαλώ να με συγχωρήσετε. Και έχω ερωτήσεις ε, που έχουν σχέση με αυτά που ελέγχθησαν ε, στην ε, Επιτροπή Κρίσης που μερικοί είπαν ότι η κρίση και το δάνειο μάλλον, το χρέος, να μοιραστεί σε όλους, να επιμεριστεί. <coughs> Για τρία χρόνια υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα και μετά από τρία χρόνια θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο ενδεχομένω ε, θα πρέπει να γίνει αυτή η αντιμετώπιση κρίσης μόνιμη και από εκεί δεν είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι τα ευρωμόλογα. Αυτά λοιπόν τα τρία χρόνια και τα απαραίτητα μέτρα πώς τα κρίνετε εσείς και κατά δεύτερον εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει αναγκαστικά να υπάρξει εναρμόνιση και σε άλλους τομείς ε, παραδείγματο χάρη ε, στο όριο συνταξιοδότηση, ε, στην κοινωνική πολιτική ή στην, στον στη φορολόγηση επιχειρήσεων στην Ιρλανδία όπου προκύπτει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Άρα δηλαδή δεν καταλήγετε κι εσείς στο ότι αυτή η κρίση ορισμένων κρατών μελών, ίσως όπως όλες οι κρίσεις ε, στην μέχρι τώρα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προκαλέσουν μια νέα πολιτική όπου θα είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παραμείνει με έναν εξάρτητη αλλά τα κράτη εκ των υστέρων να λαμβάνουν νέα μέτρα για τα οποία μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανεξάρτητη, ουσιαστικά ανεξάρτητη και εμεί θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας, τα οποία όπως σας είπα είναι πάρα πολύ απλά. Όλοι φέρουμε ευθύνη, εμείς ε, προσφέρουμε τη σταθερότητα των τιμών, το κάναμε αυτό κατά το παρελθόν, θα το κάνουμε και στο μέλλον και εσείς πρέπει να προσφέρεται αυτό που σημαίνει για μια χώρα το να είναι κράτος μέλος της κοινή αγοράς και να έχει ενιαίο νόμισμα. Κατά το παρελθόν, δυστυχώς ήμασταν φωνή βόντος εν τη τώρα όμως βλέπουμε τι προέκυψε. Βιώνουμε τη μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεν ξέρω τι άλλο μπορώ άραγε να προσθέσω. Αυτή η ιδέα του να έχουμε ευρωομόλογα, αν αυτά έχουν ως στόχο το να χρηματοδοτήσουν τον προπολογισμό των κρατών μελών, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Ανέκαθεν ήμασταν αντίθετοι σε κάτι τέτοιο. Δεν ε, λέω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να χρηματοδοτείται ή να χρηματοδοτηθεί ένα ταμείο σταθερότητας ελέγχθη αυτό πρόσφατα, σε κάποιο βαθμό οι ίδιες οι ε, καλούνται να λάβουν τις ευθύνες τους και να διχειριστούν την κατάσταση. Εγώ θέλω να πω ότι το Ταμείο μπορεί να υπάρχει για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και θα μπορεί να αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα θέματα. Αυτό που έχετε κατά νου είναι ότι μετά από τρία 3,5 χρόνια θα εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα, ίσως και νέα προβλήματα, τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Θα δείξει, δεν ξέρω τι να πω, αλλά η δική μου η παραδοχή είναι ότι παρόλα αυτά πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Πρόληψη. Δέχομαι βέβαια πλήρως και απάντησα το να ξέρει κανείς εκ των προτέρων τι πρέπει να κάνει αν προκύψουν τέτοιου προβλήματα, αυτό σαφώς και είναι σημαντικό. Παναλαμβάνω λοιπόν ότι κάθε ότι όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, το ίδιο ισχύει και για την Κομισιόν και για το Συμβούλιο. Εμείς ε, πρέπει να προσφέρουμε αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εμάς και εμείς, εν πάση περιπτώσει, το κάνουμε τόσο καλά που πολλές φορές πολλοί ξεχνούν ότι εμείς προσφέρουμε σταθερότητα τιμών σε αυτή την ε, περίεργη χρονική περίοδο που διανύουμε. Η δική μας λοιπόν η θέση ίσως ε, μας ε, καθιστά ιδιαίτερα, ιδιαίτερα υπεύθυνου και ώστε να μεταφέρουμε μηνύματα και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις νομίζω ότι ε, με το πάθο σα αν όλοι είχαν το ίδιο πάθος, πολύ εύκολα θα μπορούσαν να λυθούν πολλά προβλήματα. Επόμενο ο ο κύριο Νίτρας. Πρόεδρε, έγινε λόγος ήδη για το πιθανό συντονισμό των θέσεων ε, των κρατών μελών στα συντοξιοδοτικό, για παράδειγμα. Κατά την άποψή σας, πώς εκτιμάτε τα αιτήματα ορισμένων κρατών ε, και τη συζήτηση που γίνεται στο Συμβούλιο για το ζήτημα αυτό σε ό,τι αφορά την ε, μεγαλύτερη ελαστικότητα του δημοσίου χρέους στα πλαίσια των ε, μεταφορών, των χρηματικών μεταφορών σε ανεξάρτητα συνεξοδοτικά ταμεία. Αν θυμάμαι καλά, εννέα κράτη-μέλη ζητούν να υπάρξει διαφορετική μεταχείριση του χρέους σε τέτοιες περιπτώσεις. Εσείς υποστηρίζετε τα κριτήρια της σύγκλησης. Τι άποψη λοιπόν έχετε για την πιθανή θετική απάντηση σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών στην Ευρώπη. Και μια ερώτηση ακόμα. Δεν είναι η σωστή στιγμή να ξεκινήσουμε μια σοβαρή συζήτηση για τις μελλοντικές Ε, δεσμεύσεις των ε, προϋπολογισμών των κρατών μελών. Δεσμεύσεων που σήμερα δεν έχουν κανένα, δεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, τουλάχιστον έτσι λένε οι εκθέσεις. Σωστά, πολύ σημαντικό θέμα θέσατε. Δέχομαι, δέχομαι ότι υπάρχει ένα παράδοξο στον τωρινό τρόπο υπολογισμού των συνολικών υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά το, αυτοί που έχουν την μεγαλύτερη μέσο και μακροχρόνια διάβγεια, πλήττονται λογιστικά. Πρέπει να σας εξομολογηθώ λοιπόν ότι όντως αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Ξέρω ότι η χώρα σας το θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό και δέχομαι επίσης ότι υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Ξέρετε, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το θέμα. Συμφωνώ ωστόσο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί. Διότι ο τρόπος που δουλεύουμε τώρα φαίνεται άδικος. Άδικος, απλά και μόνο σε ό,τι αφορά την εκτίμη, την αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης. Edward. Κύριε Τρισέ, δεν αμφισβητώ το ότι είναι απαραίτητο μία χώρα να ε, σταθεροποιήσει τα δημοσιονομικά της. Όμως ε, το να ζητάμε από όλες τις χώρες να πράξουν το ίδιο, αυτό μοιάζει ε, να είναι ένα είδος ε, ιδεολογίας και αυτό πραγματικά δημιουργεί προβλήματα. Έχουμε φτάσει τώρα σε μια κατάσταση όπου λέμε καλύτερα αποταμίευση ε, παρά δαπάνες. Λέμε οι περικοπές των μισθών είναι αρετοί. Μοιάζει δηλαδή σαν να λέει σε κάποιον, κανείς σε κάποιον ε, σήκωσε τα, ανέβασε ένα κουτί για να βλέπεις πάνω από το πλήθος, αλλά άμα σηκωθούν όλοι δεν βλέπει κανείς τίποτα. Η δική μου λοιπόν η ερώτηση είναι η εξής όσον αφορά στην Κεντρική Τράπεζα. Αυτή η ε, πολιτική με μη στάνταρτ μεθόδους. Είναι κατάλληλη αυτή η πολιτική γιατί αν ε, του χρόνου όλα τα κράτη λάβουν αυτά τα μέτρα λιτότητας θεωρείται ότι αυτό μπορεί να αποτελεί λύση του προβλήματος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την πολιτική μας εγώ επιβεβαιώνω ότι πράγματι την θεωρούμε ότι είναι η ενδεδειγμένη. Εμείς ε, θεωρούμε ότι Όσον αφορά στα στάνταρτ μέτρα, το τι ενδείκνυται για να υπάρχει σταθερότητα τιμών μέσω μακροπρόθεσμα και όσον αφορά τα στάνταρτ μέτρα, εκεί θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του το ότι οι αγορές δεν λειτουργούν απόλυτα σωστά. Άρα δηλαδή η νομισματική μας πολιτική πρέπει να μεταδίδεται με το σωστό τρόπο. Εμείς θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλες τις αποφάσεις που είναι απαραίτητες για να υπάρχει σταθερότητα τιμών. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες και ανεξάρτητα από τα στοιχεία που μπορούν να προκύψουν είτε μέσα είτε και έξω από την Ευρώπη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό είμαστε αξιόπιστοι γιατί οι παρατηρητές ανατρέχουν στο παρελθόν και από εκεί ορμόμενοι εξάγουν τα συμπεράσματά τους για το μέλλον. Ε, σας είπα λοιπόν, εμείς θεωρώ ότι είμαστε σωστοί στο στόχο μας. Κοντά στο 2, λίγο πιο κάτω από το 2, άρα δηλαδή με τον τρόπο αυτό δεν εμφανίζεται ούτε κίνδυνος πληθωρισμού ούτε αποπληθωρισμού. Σας λέω λοιπόν και πάλι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε πολλές περιπτώσεις πράγματι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ε, δεν διακυβεύονται μη γραμμικά μέτρα και δρομολογώντας δημοσιονομικές πολιτικές οι οποίες ε, θα είναι καθησυχαστικές μέσω πρόθεσμα, με τον τρόπο αυτό επιτυχάνει κανείς καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί σας λέω και πάλι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνη σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης είναι και θα είναι πολύ αρνητική αν δεν ληφθεί καμία απόφαση. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και όπως σας είπα όσον αφορά εμάς εμείς ε, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να ε, διασφαλίζουμε, να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε αξιόπιστη πολιτική τιμών μέσω πρόθεσμα. Ε, ανέφερα νομίζω αρκετά θέματα όσον αφορά στην ε, ε, ξελ, εξελίξεις της νομισματικές και στους μισθούς. Επιτρέψτε μου μόνο να προσθέσω ότι σήμερα το πρωί είχαμε τις εξελίξεις του M3 που είναι στο 1,1%. Ήμασταν στο 0,2% τον Ιούλιο και τον Ιούνιο και αν δούμε λιγάκι την άλλη πλευρά του M3, βλέπουμε μία μικρή αύξηση των μισθών, των δανείων, των δανείων στα νοικοκυριά και αρνητική εξέλιξη των ε, επιχειρηματικών δανείων. Βλέπουμε λοιπόν ε, ένα φαινόμενο το οποίο το αναλύσει κανείς νομισματικά καταλήγει στο ότι τελικά πράγματι προκύπτει δυναμισμός. Αυτό δεν εκπλήσει. Πάντα μετά την ύφεση εμφανίζεται αύξηση χορήγησης δανείων πρώτα στα νοικοκυριά και μετά στις επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε κατ' ουσίαν ε, το είχαμε προβλέψει. Βεβαίως οφείλουμε να το ομολογήσουμε ότι είχαμε ε, δυστυχώς μια πολύ έντονη ύφεση. Τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Τρισέ για τα σχόλιά του στο ξεκίνημα για την βιώσιμη οικονομία και τα κίνητρα προς τα κράτη-μέλη για τη διαχείριση των έρηματων. Εγώ θα θα για τις κυρώσεις. Αν κάποιος πολίτης έχει προβλήματα, θα πρέπει να διαχειριστεί όχι μόνο τις δαπάνες, αλλά και το χρέος του περιορίζοντας ε, τις πιστοτικές κάρτες κλπ. Όταν μια χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη προτείνουν μεγάλα πρόστιμα. Άλλοι προτείνουν την παρακράτηση πόρων. Με άλλα λόγια, μείωση των κονδυλίων για τη συγκεκριμένη χώρα στη στιγμή που το χρειάζεται. Κοιτάζω επίσης και τα επιτόκια και το περίπλοκο σύστημα της εγκυοδοσίας των ευρωπαϊκών, ε, του, Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοδότησης και την, το υψηλό κόστος δανεισμού. Ο συνδυασμός υψηλών προστήμων, υψηλών επιτοκίων και υψηλών και υψηλού κόστου δανεισμού δίνουμε στα κράτη-μέλη μια ακριβή ψηλή πιστοτική κάρτα, μειώνοντας τις δυνατότητές τους να ελέγξουν το έλλειμμά του. Ευχαριστώ. Δεν εκπλήσει βέβαια το ότι όταν ε, συμπεριφέρεσαι λάθος πρέπει να πληρώσεις ένα κάποιο τίμημα. Αυτό είναι σαφές. Και το γεγονός ότι η ίδια η βοήθεια έρχεται με ένα τίμημα υψηλότερο προέρχεται από τους εταίρους σου, τις άλλες κυβερνήσεις που λένε ότι δεν μπορούμε να βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση που να δημιουργήσουμε χαμηλότερο κίνδυνο γιατί θα πρέπει να παρέμβουμε εμείς και να σας βοηθήσουμε. Άρα να μην έχεις κίνητρο. Πάντα λοιπόν η κατάσταση είναι λεπτή. Υπάρχει λογική σε αυτό που γίνεται, δεν μπορώ να σας πω ότι θα έπρεπε να δράσουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Οι καταστάσεις αυτές δεν πρέπει να εμφανίζονται, πρέπει να τις αποφεύγουμε. Και ο ηθικός αυτός κίνδυνος είναι κάτι που δείχνει ότι το, το βλέπει και το κάθε κοινοβούλιο και εσείς και όλοι, με ευθύνη κιόλα, με υπευθυνότητα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, ευχαριστώ και ε, για τις ερωτήσεις του συναδέλφου τις οποίες δόθηκαν με πάθος απαντήσεις. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι στο τέλος Νοεμβρίου στις 4.30 το απόγευμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσουμε εμείς τώρα σε λίγη ώρα όμως. Κάνουμε μια μικρή διακοπή. Okay, those who are leaving could do so quickly and quietly. Uh, then we can uh, proceed. Καλώς. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Είναι το σημείο 6. Η βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ. Θα έχουμε μια συζήτηση για τις τροπολογίες στην έκθεση ΦΕΙΟ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Φέιο, θα ήθελα να ζητήσω από αυτούς οι οποίοι μιλούν να βγουν από την αίθουσα, γιατί ο κύριος Φέιο θα πρέπει να μας δώσει εξηγήσεις για το τι θα γίνει με τις σημαντικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στην έκθεσή του. Um, I can, do what they do in the House of Commons and start naming Μπορούσα να κάνω αυτό το οποίο γίνεται στην κάτω βουλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, να ονοματίζω τους βουλευτές που είναι άτακτοι. Λοιπόν, κύριε Φέγιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Η έκθεση για την οικονομική διακυβέρνηση της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σταθερότητας ε, της ζώνης ευρώ προκάλεσαν 254 τροπολογίες. E Ευχαριστώ τις διάφορες πολιτικές ομάδες οι οποίες ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα γύρω από την έκθεσή μου και κατέθεσαν και τις ιδέες τους μέσω των τροπολογιών. Θα ήθελα σαν εισηγητής να ομολογήσω για μια ακόμη φορά ότι είμαι πλήρως διαθέσιμος να ακούσω τους συναδέλφους και τις τροπολογίες τους. Έχω ήδη έρθει σε επαφή και με τους σκιώδεις εισηγητές και θα ήθελα να πω στα μέλη επίσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ότι είμαι απόλυτα διαθέσιμος να προχωρήσουμε σε διάλογο μαζί τους. Έχουμε διαπιστώσει και σε άλλες συζητήσεις ε, που έχουν προηγηθεί. Η έκθεση περιλαμβάνει οκτώ βασικές συστάσεις. Οι δύο από τις συστάσεις αυτές έχουν γίνει αντικείμενο πολλαπλών τροπολογιών. Καταρχάς, το εποπτικό πλαίσιο της μακροοικονομικής εξέλιξης στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη. Το δεύτερο θέμα αφορά την ενίσχυση του ε, Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα ήθελα και για τις δύο αυτές περιπτώσεις να πω ότι ιδιαίτερα σε σχέση με τον λεγόμενο πολυμερή έλεγχο, οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί σχετικά με τους δείκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Να πω εδώ ότι οι δείκτες αυτοί είναι απαραίτητοι εφόσον θέλουμε να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος και εποπτεία και εφόσον θέλουμε να αυξήσουμε ε, τα επίπεδα σταθερότητας. Υπάρχουν κανόνες λοιπόν που αφορούν τον έλεγχο του χρέους και να διευκρινίσω εδώ ότι η έκθεση λαμβάνει υπόψη το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Υπάρχουν ορισμένε ιδέες οι οποίες έχουν κατατεθεί και για τις θεσμικές μελλοντικέ εξελίξεις, αλλά δεν είναι αυτό το αντικείμενο. Επίσης προτείνονται διάφορες ιδέες για ευρωομόλογα. Ευρωομόλογα τα οποία θα ε, προκαλέσουν, θα έλεγα, κάποιες αλλαγές στη συνθήκη εφόσον γίνουν δεκτά σαν ιδέα θα πρέπει να τα μελετήσουμε αυτά σε μια ιστερότερη φάση και θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες έχουμε στο μέλλον να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες στη συνθήκη αλλαγές. Το βασικό πάντως πλαίσιο της συνθήκης της συγκεκριμένη αφορά τη λεγόμενη δευτερογενή νομοθεσία. Αυτή δηλαδή η οποία μπορεί να προχωρήσει και να εφαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες νόμους. Επ' αυτού υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μέσω των τροπολογιών. Καταρχάς υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τις εξαιρέσεις. Αυτό ισχύει επίσης και για τις συγκεκριμένες διαδικασίες για το δημόσιο χρέος και για τον σεβασμό του 60% του ΑΕΠ σχετικά με το δημόσιο χρέος. Γύρω από όλα αυτά ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία στα οποία θα καταλήξουμε για να ορίσουμε σωστά το πλαίσιο εποπτείας. Η έκθεσή μου λοιπόν νομίζω ότι αντικατοπτρίζει μια ισχυρή μεν αλλά και συνενετική άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περιλαμβάνει από τη μία κάποια καινοτόμα στοιχεία τα οποία έχουν προταθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή και από την άλλη δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προχωρήσει ε, στις σχέσεις του με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να προσθέσω ότι είμαι <clears throat> διαθέσιμος να δεχτώ τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί Είμαι ανοιχτός στον διάλογο και να προσθέσω ακόμα ότι η συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει θα είναι για μένα μια συζήτηση η οποία δεν θα μπορεί παρά να βελτιώσει τις λύσεις οι οποίες έχουν μέχρι τώρα προταθεί όπως αυτές περιλαμβάνονται στην έκθεσή μου. Τελειώνοντας, λέει ο κύριος Φέιο, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω και το λέω αυτό πολύ σοβαρά, Ελπίζω λοιπόν ότι όταν στις 5 Οκτωβρίου ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη έκθεση τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά και θα ήθελα να συνεχιστεί η στενή μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Αυτό που προτείνω είναι να ακούσουμε τους σκιώδεις και κατόπιν τους υπόλοιπους Αγωγητές. Ελίζα, πρώτη. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα αγγλικά για να μιλήσω γρηγορότερα. Ξεκινώ εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου προς τον κύριο Φέιο. Είχε ένα πολύ ανοιχτό πνεύμα συμβιβασμού και εγώ πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο σε μια τόσο κρίσιμη και ευαίσθητη ομάδα θεμάτων θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να έχουμε μια κοινή θέση. Με αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο εξ ονόματος ε, της ομάδας των σοσιαλιστών και δημοκρατών υπέβαλα πολλές τροπολογίες και ξεκίνω έναν πολύ στενό διάλογο με τον κύριο Φέιο το ΕΛΚ γενικότερα, τους φιλελεύθερους και τις υπόλοιπες ομάδες στο πλαίσιο των τροπολογιών. Από πλευράς μου θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να μπούμε σε ένα πνεύμα συμβιβαστικής προσέγγισης. Όπως είπε ο κύριος Φέιο, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια γενικευμένη ευρεία συμφωνία για τις συστάσεις από τον αριθμό 3 στον αριθμό 8. Ωστόσο, θεωρώ παρά τα σημαντικό να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Μία από αυτές είναι ο τύπος του εγγράφου και της έκθεσης, ακολουθώντας το άρθρο 42. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς όταν ζητούμε συγκεκριμένα πράγματα από την Επιτροπή και στο συγκεκριμένο αυτό κλάδο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν ζητούμε να υπάρξει για παράδειγμα μια ομάδα υψηλού επίπεδου ή να εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημιουργίας Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, κάτι επί το οποίο συμφωνούμε όλοι, να δίνουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ένα χρονοδιάγραμμα για να κάνει το συγκεκριμένο έργο επιτροπή, ιδίω όταν μιλούμε για να υπάρξει μια σειρά εκθέσεων βιωσιμότητες για το τι θέλουμε να υλοποιηθεί κατόπιν. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας τις συστάσεις του Κοινοβουλίου για το προσωπικό του Eurogroup. Εδώ υπάρχουν πολλές προτάσει τροπολογία. Εμείς έχουμε μια πρόταση που ζητά να αναλυθεί το τι θα γίνει με, την, με το προσωπικό του Eurogroup σε συνδυασμό με την εξωτερική ημερήσια διάταξη της ε, ε, ε, Ένωση, δηλαδή τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ένωση που είναι επικεφαλή των εξωτερικών υποθέσεων. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να μπούμε σε μια ουσιαστική συζήτηση για το πού θέλουμε να προχωρήσουμε. Βεβαίω είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για να ενισχύσουμε και να καταστήσουμε αποτελεσματικότερη τη διαχείριση του Eurogroup. Αυτό για τις τροπολογίες, για τις συστάσεις, συγγνώμη, 3 έως 8. Τώρα, κάτι άλλο για τα, τις συστάσεις 1 και 2. Εδώ συμφωνώ, τα προβλήματα είναι πιο σύνθετα. Και ένα από τα ζητήματα που το Κοινοβούλιο, εμείς ιδιαίτερα στην Επιτροπή πρέπει να συζητήσουμε, είναι μέχρι πού θα φτάσουμε διαχωρίζοντας τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσει για το Eurogroup και το τι γίνεται με τους υπόλοιπους, την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συνολικά. Αναγνωρίζω ότι πολλές τροπολογίες ε, της κυρίας Φόρντ υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα να διαχωρίζεται πάντα η, το Eurogroup από τους υπόλοιπους. Κατά την άποψή μου, οι υποχρεώσεις για τις χώρες του Eurogroup είναι αυτονόητες. Το πρόβλημα είναι πώς θα διαχειριστούμε τη σχέση μεταξύ των χωρών του Eurogroup και των υπόλοιπων χωρών της Ένωσης. Λαμβάνοντα υπόψη ότι πολλές από τις χώρες αυτές δεν είναι ακόμα μέλη του Eurogroup που προετοιμάζονται ωστόσο για ένταξή τους στη ζώνη του ευρώ. Πώς λοιπόν μπορεί να ζητήσεις καταρχήν από αυτές να μην αυξηθεί η δυνατότητα του να επιλέγεις τι θες και τι δεν θες αλλά μέσα ή έξω από την ε, Ευρωζώνη αλλά να αναγνωρίζεις τις υποχρεώσεις που είναι κοινέ είτε είσαι μέσα είτε είσαι έξω από την Ευρωζώνη. Αυτά τα θέματα νομίζω πρέπει να τα δούμε. Δεύτερο ζήτημα. Λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν είναι εδώ η κυρία Χούπνερ. Η συμβιβαστική 10α είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί προσπαθεί να προβλέψει τον αντίκτυπο που θα έχει μία χώρα στην άλλη. Αλλά λέει εκεί το κείμενο ότι πρέπει να υπάρχουν κατόφλια, να δημιουργήσει κατόφλια η Επιτροπή. Τεχνικά αυτό είναι εφικτό. Δεν το ξέρω. Έχω λοιπόν κάποια προβλήματα με αυτή την πρόταση συμβιβασμού. Τώρα, έλλειμμα χρέος. Είναι σαφές ότι τα κριτήρια του χρέους και τα κριτήρια του ελλείμματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο ενιαίο τρόπο. Διότι ε, είναι ένα από τα προβλήματα του συμφώνου. Από τη μια μεριά δίνει μεγάλη έμφαση στα κριτήρια του ελλείμματος, αλλά όχι αρκετή στα κριτήρια του χρέους. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον αυτοματισμό 60% χρέος αυτόματα να δημιουργεί κυρώσεις ή να ξεκινούν συστάσεις. Πρέπει να ξέρουμε καλύτερα πώς συσχετίζεται χρέος και έλλειμμα, πώς συνδέονται μεταξύ τους, να μην δημιουργούμε νούμερα 3% από εδώ, 60% από εκεί. Γιατί ακριβώς ο συνδυασμός τους επιτρέπει να καταλάβουμε πώς είναι η εξέλιξη των δύο. Και να μην έχουμε όρια. Πρακτικά λοιπόν και τεχνικά δεν θεωρώ ότι τα όρια αυτά πρέπει να είναι αυτόματα. Είναι, δεν, έχουν, δεν έχει νόημα. Κάτι πιο σημαντικό και πολιτικά εξαιρετικά ευαίσθητο νομίζω. Πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε στις ήμι ε, ή ονή αυτόματες κυρώσεις που προτείνει η αυτοματες κυρωσεις που προτεινει επιτροπη χωρις να περάσουμε από το Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο ζήτημα. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ κάποιων μεγάλων ομάδων για την Επιτροπή Αντιμετώπισης της Κρίσης πρέπει να έχει μία ισορροπημένη γλώσσα, να ενισχύσουμε τις ε, αρμοδιότητες της Επιτροπής, αλλά όχι να τις αγνοήσουμε, να αγνοήσουμε παντελή, παντελώς τις ε, ε, γραμμές του Συμβουλίου, διότι ε, κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας. Συνέβη κάτι τέτοιο στο παρελθόν και νομίζω ότι δεν θα λειτουργήσει να υπάρχουν κυρώσεις της Κομισιόν ε, σε κάποιους χώρες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα λόγου των κυβερνήσεων. Λοιπόν, ναι, η, τοπο, η επιβολή κυρώσεων να είναι υπό την καθαρή καθοδήγη της Επιτροπής, όχι όμως ένας αυτόματος ε, τρόπος επιβολής κυρώσεων σε κυρίαρχες χώρες από την Επιτροπή χωρίς λόγο του Συμβουλίου. Τελευταία παρατήρηση. Η ερμηνεία της οικονομικής διακυβέρνησης έγινε στην πράξη ως ενίσχυση του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Η ιδέα που υποκρύπτεται το πίσω από την οικονομική διακυβέρνηση ήταν να περισσότερο να εισαχθεί παράλληλα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξης και ένα ταυτόχρονα τμήμα απασχόλησης. Γιατί στην πραγματικότητα το σύμφωνο έγινε σύμφωνο σταθερότητας αλλά όχι ανάπτυξης. Λόγω του ότι ακριβώς ε, η προσπάθεια σταθερότητας έγινε εις βάρος της ανάπτυξης υπήρξαν αποκλήσεις των οικονομιών και άρα μείωση της απασχόλησης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συγκεκριμένη σύσταση που να λέει ότι σε κάθε χώρα θα πρέπει το σύμφωνο σταθερότητας και απασχόλησης να υποκαταστήσει το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο, σημαντικό ζήτημα για την πολιτική μου ομάδα και ευχαριστώ τις ε, διάφορες πλευρές, θα παρακαλούσα μάλλον τις διάφορες πλευρές να βρούμε μια κοινή γλώσσα σε αυτό το ζήτημα. για το μέλλον της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ. Ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας. Να υπογραμμίσω εκ νέου ότι βρισκόμαστε σε τροχιά συμφωνίας. Ελπίζω να βρεθούμε σε μια κοινή θέση γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα μιλήσω στα ισπανικά για να, γιατί ε, καταλαβαίνόμαστε με τον κύριο Φέιο και έτσι δεν θα μιλήσω αγγλικά. Υπέβαλα 30 τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης, πολλές από τις οποίες υπογράφηκαν και από τους συναδέλφους της φιλελεύθερης ομάδας. Μέχρι τώρα 15 από αυτές τις περιέλαβε ο κύριος Φέγιος στα συμβαστικά κείμενα του. Ελπίζω λοιπόν μέχρι το τέλος να τον πείσω ότι και άλλε δικές μου τρομολογίε ε, είναι καλό να μπουν στο συμβαστή, στις, συμβαστικέ συμβαστικές τοπολογίες Πάντως, να πω τέσσερα σημαντικά θέματα για μένα. Πρώτον, συμφωνώ με τη σκληρή θέση των φιλελεύθερων. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος των χωρών που μπαίνουν στη ζώνη ευρώ, ούτω ώστε να τηρούν τις δεσμεύσεις του συμφώνου. Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα και το χρέος. Στην περίπτωσή μου, την ισπανική περίπτωση, το ε, χρέος αυξάνεται σημαντικά και αποτελεί πλέον ένα διαρθρωτικό ζήτημα. Πολύ σημαντικό αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ. Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί και αυστηροί με τις χώρες που μπαίνουν στη ζώνη, με τις χώρες της Ευρωζώνης απαιτώντα μία πειθαρχία. Η Ισπανία δεν είχε σκανδιναβική συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό. Ιδίω με τους σοσιαλιστές. Τέλο πάντων, συγγνώμη ζητώ από του συναδέλφου, αυτή είναι η άποψή μου. Πάντω, θεωρώ σημαντικό το ότι υπάρχει σαφή δέσμευση για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Την περασμένη Τετάρτη στο Στρασβούργο είχαμε ένα γεύμα με τον Άξελ Βέμπερ, κάποιοι βουλευτέ, ο οποίο ε, μίλησε τελείως, ήταν αντίθετο τελείως αντίθετος με μια τέτοια ιδέα. Πάντω είναι θετικό να υπάρχει σαφή θέση του Κοινοβουλίου για το κατά πόσο πρέπει η Ένωση να έχει ή όχι έναν μηχανισμό ταχεία απάντηση, δικό τη μηχανισμό, σε τέτοιε κρίσει και να μην περιμένει από διεθνεί ε, οργανισμούς. θεωρώ θετικό, θετική την αναφορά στην έκδοση ευρωμολόγων. και την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην κατά προτεραιότητα χρησιμοποίηση των ομολόγων αυτών σε ευρωπαϊκά έργα υποδομών. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η Ισπανία δεν έχει συνδρομική σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Υπάρχουν όχι μόνο κανονιστικά, αλλά και φυσικά εμπόδια, η διαφορά ε, εύρους γραμμής ε, που εμποδίζουν την σύνδεση της Ισπανίας, του σιδηροδρομικού συστήματος της Ισπανίας με το ευρωπαϊκό. Να κάτι που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τα ευρωομόλογα. Επίσης, η, μια τροπολογία μου, η 224, ζητά από την Επιτροπή να διεξάγει μια μελέτη για τα υπέρ και τα κατά και τις δυνατότητες δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κοινού ε, λογιστήριου του κράτους. Είχα, όταν μιλούσα με ψηφοφόρους μου, με ρωτούσαν τι θα πει η οικονομική διακυβέρνηση, τι σημαίνει. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να αποκτήσει μια πραγματική οικονομική κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή η Ένωση είναι μια Ένωση ανεξαρτήτων κρατών. Έχουμε ένα κοινό νόμισμα, έχουμε μια κοινή νομισματική πολιτική, αλλά δεν έχουμε σχεδόν καθόλου ε, δημοσιονομική εναρμόνιση και χωρίς να έχουμε ένα κοινό ουσιαστικό προϋπολογισμό δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Χαίρο διότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το διάλογο με τον κύριο Φαϊό και ελπίζω να υποβάλουμε να υποβάλει ο, ο, ο συντάξη μια σειρά συμβαστικών προτάσεων που θα καλύπτουν και τι δικέ μα θέσει. Βίκη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον ε, κύριο Φαϊό. Άκουσα πολύ προσεκτικά, που άκουσε πολύ προσεκτικά τις ανησυχίες μας κατέθεσα τροπολογίες ε, και αναφέρω ε, πού θα πρέπει να έχουμε την Ευρωζώνη και πού ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες, να δούμε πού λειτουργεί και πού όχι. Και αυτό για να παραμείνουμε σε κάποιο βαθμό μέσα στο σύμφωνο σταθερότητας στη δική μου τη χώρα, αλλά και σε άλλες υπάρχουν ανησυχίε. Μερικοί ε, θέλουν ίσως να αλλάξει το σύμφωνο σταθερότητας. Εγώ έχω καταθέσει σχετική ε, τροπολογία γιατί ίσως στο μέλλον θα έπρεπε να σκεφτούμε λιγάκι την αλλαγή του σύμφωνου σταθερότητας και ε, θα πρέπει ίσως να το έχουμε κατά νου. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό η έκθεση αυτή να παραμείνει επί της ουσίας. Παραδείγματος χάρη, βλέποντας τους δείκτες, τι πρέπει να προσμετράτε και τι όχι στο μέλλον. Ας ε, δούμε τους δείκτες και ας παραμείνουμε επί της ουσίας στο πώς ε, η σταθερότητα να λειτουργεί στο μέλλον και όχι σε τελική ανάλυση να ε, συγχέονται τα πράγματα. Ας παραμείνουμε ξεκάθαροι. Όσον αφορά το θέμα των προστήμων, είπα ήδη ότι υπάρχει μεγάλη ευαισθησία, ότι με τα πρόστιμα κατ' ουσίαν ε, δίνουμε την, ε, το τελικό χτύπημα. Κάποιος που είναι πληγωμένος το χτυπάμε μέχρι θανάτου. Ε, πρέπει λοιπόν να προσέξουμε έτσι ώστε η συζήτηση να μην εκτροχιαστεί πλήρως. Τώρα, μία πρόταση ότι ίσως αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε τους προπολογισμού των κρατών μελών με ένα είδος stress test. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που μια κυβέρνηση έχει ε, αρνητικές εξελίξεις στον προπολογισμό, οι αγορές λαμβάνουν τα μέτρα τους. Και όταν ένας υπουργό Οικονομικών κάνει τις προβλέψεις του, ε, αρχίζει αυτομάτως η συζήτηση. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, τράπεζες. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσω προσεκτικά τα επιχειρήματα των άλλων, των υπολείπων. Κατά τη δική μου άποψη είναι απόλυτα σαφές ότι η ευθύνη για τους εθνικούς προπολογισμούς παραμένει στις εθνικές κυβερνήσεις. Και κατανοώ βέβαια ε, τα ωφέλη που θα προκύψουν από το ευρωπαϊκό εξάμεινο για να έχουμε ε, σωστές προβλέψεις και να δούμε τις επιπτώσεις ε, σε άλλα κρατημέλη, αλλά τελικά η ευθύνη παραμένει σε εθνικές κυβερνήσεις και ευχαριστώ που ε, δεχθήκατε την ε, ε, τροπολογία που δείχνει ότι σέβεστε τις κοινοβουλευτικές προθεσμίες. Ορισμένα κρατημέλη, κυρίως που κάθονται από αυτή την πλευρά, επιθυμούν η Κομισιό να κοιτάει τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα. Εμείς όμως θέλουμε να δούμε και τις προτεραιότητες δαπανών των κρατών μελών. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ προχωρημένο. Ε, για μένα τουλάχιστον, εφόσον ένα κράτος μέλος καταρτίζει τον προπολογισμό του με συνετό τρόπο, θα πρέπει το ίδιο το κράτος να μπορεί να αποφασίζει ε, πώς θα ε, δαπανίσει τα κονδύλια του και όχι να του επιβάλλει η Ευρώπη το τι θα πρέπει να εκταμιεύσει για την υγεία ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, οι κυρώσεις για να μην μπορούν τα κράτη-μέλη να παίρνουν χρήματα από τα διευθυντικά ταμεία. Επ' αυτού μου αρέσουν οι παρατηρήσει του ε, Βόλφ. Όσον αφορά τα ευρωμόλογα, ε, θα μου άρεσε βέβαια πάρα πολύ να βρεθεί ένας φτηνός τρόπος ε, δανεισμού. Αυτό θα ήταν θαυμάσιο, αλλά νομίζω όμως ότι αυτό ενέχει πολλούς ηθικούς κινδύνους. Ε, κοινή εγγύηση από 27 κράτη-μέλη χώρες της Ευρωζώνης που να πληρώσει, να ε, εγγυηθεί για ε, τους συνδρόμους ε, στην Ισπανία. Αν όμως μία ένα κράτος κηρύξει στάση πληρωμών, χρεοκοπία, αυτομάτως καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στους συνδρόμους της Ισπανίας. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν η κίνδυνη από αυτό που πιστεύετε εσείς ως κοινή ευθύνη για την διαχείριση των προϋπολογισμών. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί να έχει πολύ περισσότερους κινδύνους από αυτούς που φανταζόμαστε. Τώρα, για την τροπολογία που κατέθεσε η Πρόεδρος όσον αφορά τους ε, μηχανισμούς ε, για την αντιμετώπιση των χρεών, υπάρχει μια θαυμάσια μελέτη που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα το Κοινοβούλιο επί του θέματος και έχει να κάνει με το ότι οι τράπεζες μπορούν να αγοράσουν τα δάνεια χωρίς να πρέπει να παρακρατήσουν και ε, κεφάλαια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Αυτή την, ε, τον μηδενικό κίνδυνο στην αξιολόγηση κυρίως για τις χώρες της Ευρωζώνης. Αν θέλει κανείς ε, να μην ε, έχει κανένα κίνδυνο στο να εκδώσει χρήμα, θα πρέπει στην αξιολόγηση να είναι μηδενικού κινδύνου. Ο Φιλίπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Διώργο για την έκθεσή του και ιδιαίτερα για την αποδοχή των συνενετικών προτάσεων θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μου μπορεί να συμφωνήσει με τις περισσότερες από τις προτάσεις αυτές. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, ιδιαίτερα στο θέμα της φορολογίας. Είναι ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε με πολύ προσεκτικό τρόπο στην τροπολογία μας. Όταν μιλάμε για υποστηρίξιμες οικονομικές ή δημοσιονομικές μάλλον ρυθμίσεις, θα πρέπει να είναι αντίστοιχα και τα έσοδα και φυσικά και οι δαπάνες. Θα θέλαμε λοιπόν λίγο περισσότερο αυτά να τα δούμε στην έκθεση χωρίς να μπαίνουμε σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχουν όμως ορισμένα θέματα τα οποία τίθενται σε τακτική συζήτηση όπως η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, το CCCTB, Νομίζω ότι όλα αυτά είναι θέματα στα οποία μπορεί να υπάρξει μια αναφορά. Σχετικά τώρα με αυτά τα οποία δεν καλύπτονται από τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Αυτά τα σημεία εσείς πιστεύετε ότι δεν θα πρέπει να ανήκουν στην έκθεση πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα να θέσω δύο επιπλέον σημεία. Το ένα αναφέρεται στην να είναι πραγματικά υποστηρίξιμες ε, οι μακροοικονομικές μας πολιτικές. Σε αυτές τις πολιτικές ε, θα πρέπει να υπάρχει σωστή, αν θέλουμε, παράλληλη πορεία ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει επίσης το θέμα ε, των... Ξέρουμε ότι το πλεόνασμα του ενός είναι το έλλειμμα του άλλου σε ορισμένες περιπτώσεις. Και όταν πρέπει να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης υπερβολικών ελλημάτων. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και με τα υπερβολικά πλεονάσματα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις δύο αυτές περιπτώσεις με ισορροπία. Για τη διαδικασία τώρα. Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιο παραλληλισμό εδώ, να κάνουμε κάποιο παραλληλισμό και με άλλες εκθέσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα στο οποίο έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Πρέπει να τελειώνουμε με την έκθεση αυτή και να ξεκινήσουμε τη δουλειά πάρα πολύ σύντομα επί της ουσίας θα πρέπει να ξεμπερδεύουμε σε εισαγωγικά θα έλεγα γιατί νομίζω ότι μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα, Σύντομα ο σκιώδης εισηγητής μας είναι ο Ραμών. Στα πλαίσια της προοπτικής των κειμένων που μας αναμένουν. Ευχαριστώ τον Διόγο για τον δεκτικό τρόπο με τον οποίο μας αντιμετώπισε να πούμε τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα. Την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κυκλοφορήσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Υπάρχει η Task Force Van Rompuy, η οποία σίγουρα μπορεί να δώσει κάποιες ιδέες, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα της πρωτοβουλίας στη συγκεκριμένη περίπτωση και εμείς φυσικά συνεισφέρουμε στη συζήτηση. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να υιοθετήσουμε την έκθεση αυτή γρήγορα, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Θα πρέπει να δούμε επίσης τι γίνεται με τις επιμέρους προτάσεις. Η προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε για το πακέτο είναι μια προσπάθεια η οποία έχει σαν στόχο να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια ανάμεσα στα μέτρα τα οποία μπορούμε τώρα να προτείνουμε στα πλαίσια των συνθήκων σε κάποια μέτρα τα οποία ξεπερνούν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση για την εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ. Και εδώ επανέρχομαι στην ερώτηση του Λάμπερτς. Πιστεύετε ότι υπάρχει λόγος να το συμπεριλάβουμε το θέμα αυτό. Εγώ θέλω ε, να επαναλάβουμε το αίτημα προς το Συμβούλιο μιας εκπροσώπησης της ζώνης ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ιδιαίτερα και με τα αιτήματα των αναδειωμένων χωρών οικονομιών που ζητούν τη δική τους θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί συντονισμένα. Όπως ακριβώς το κάναμε ε, και για τη δημιουργία του ευρώ με ένα χρονοδιάγραμμα πολύ συγκεκριμένο. Έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλη σημασία και γι' αυτό εγώ έκανα τροπολογίε για τη γραμματεία του Eurogroup. Δεν πρέπει να ενισχύουμε ιδιαίτερα τι δομέ του Συμβουλίου που δημιουργούν συγχύσει. Δεν θα ήθελα να κάνω άλλα σχόλια για την Task Force. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα δώσει. Έχω πολλέ επιφυλάξει. Ό,τι όμω έχει στόχο τη διευκρίνηση των αρμοδιοτήτων και την προσφυγή στην κοινοτική μέθοδο είναι κάτι το θετικό. Και εδώ φτάνω στην τελευταία μου παρατήρηση. Ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου μέσα σε όλα αυτά. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον ε, επαναλαμβάνουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες. Να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ρόλο της ένα εποπτικό ρόλο, αυξημένο. Να υπάρξει εκμετάλλευση της εμπειρογνωμοσύνης για τον συστημικό κίνδυνο και για τις νέες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά ο ρόλος του Κοινοβουλίου ποιος είναι. Εγώ είμαι υπέρ ανεξάρτητων αρχών, ευρωπαϊκών αρχών, οι οποίες όμως να έχουν και μια κάποια ευθύνη μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι μπορούμε να προτείνουμε το έξυπνο, το αποτελεσματικό, έτσι ώστε όταν υπάρχει ρήξη της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη-μέλη, να μπορέσουμε χωρίς ταμπού, χωρίς ε, να θέλουμε να προχωρήσουμε σε κυνήγι μαγισσών, Πώς να μπορέσουμε να κάνουμε όμως μια συζήτηση δημόσια και υπερεθνική χωρίς ε, ε, περιορισμούς. Αυτό είναι το κοινοβούλιο. Και ε, νομίζω ότι εφόσον θέλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις προβλέψεις της συνθήκης, γιατί είναι μια κοινή ευθύνη το να υπάρχει ένα κοινό νόμισμα, και Βίκυ, συγγνώμη, αλλά τα κοινοβούλια των κρατών μελών α κάνουν τη δουλειά του. Εγώ δεν έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο με τον οποίο τα κοινοβούλια των κρατών μελών παραβίασαν επανειλημμένα τις υποχρεώσεις που έχουν επικυρώσει συγκεκριμένες χώρες με πολύ συγκεκριμένε ε, ευθύνε και συνέπειε για χώρε όπω η δική μου. Λοιπόν, ναι, αλλά και οι, τα εθνικά κοινοβούλια να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Έχουν δικαίως τους νέες ευθύνες με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ας τις ασκήσουν επιτέλους. Επειδή είναι ήδη αργά, θα ήθελα να κάνω ένα ε, σχόλιο επί της διαδικασίας. Εγώ νομίζω το εξής. Το κατά πόσον τελικά θα μπορέσουμε να έχουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή πρόταση επί του θέματος, νομίζω ότι αυτό θα είναι καθοριστική σημασίας για την ικανότητα του Κοινοβουλίου να παίξει σημαντικό ρόλο. Στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παίξαμε σημαντικό ρόλο σε όλες τις εκθέσεις και επικρατεί η άποψη ότι αυτό βοήθησε στο να γίνουν οι προτάσεις καλύτερες για τους πολίτες και επίσης ε, βελτίωσε και τις ε, προτάσεις αν τις αναλύσει κανείς χωρίς ε, ιδεολογικές προκαταλήψεις. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον θα μπορέσουμε τελικά στην δική μας την Επιτροπή να παίξουμε σημαντικό ρόλο στο να υπάρχει μια ουσιαστική ευρωπαϊκή προοπτική. Ε, παίρνω λοιπόν πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που είπε η συνάδελφός μου η Ελίζα. το είπαν και άλλοι τα πράγματα δεν είναι πιο δύσκολα. Τα είδαμε και σε κάποιες συζητήσεις που έγινε στην Επιτροπή Κρίσης. Ο κύριος Φέιο έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει και νομίζω και το σύνολο της Επιτροπής επίσης, διότι αν σε ορισμένα θέματα κλειδί σε αυτήν την έκθεση ψηφίσουμε με τον παραδοσιακό τρόπο για μακροοικονομικά θέματα, τότε τελικά θα αποδυναμώσουμε μια ισχυρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι το οποίο μας τελικά χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε όταν θα μπούμε στα πραγματικά προβλήματα, όταν θα αρχίσουμε να συζητάμε με το Συμβούλιο, το οποίο δεν είναι πρόθυμο να ε, εξετάσει ισχυρές, ουσιαστικές ε, ευρωπαϊκές προοπτικές. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, να λάβουν αυτό το θέμα σοβαρά υπόψη τους. Το θέμα δεν είναι να κερδίσει κανείς τη μία την άλλη ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Αυτό που παίζει ρόλο είναι να επιτύχουμε λύσεις οι οποίες θα γεφυρώνουν τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην αποκαλούμενη αριστερά και την αποκαλούμενη δεξιά. Και αυτό για να επιτύχουμε μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση στο Συμβούλιο. Αυτό ήθελα να πω και προσβλέπω ε, στην ε, συνεισφορά όλων των συναδέλφων που εργάστηκαν τους τελευταίους μήνες για αυτή την κοινή γραμμή. Γιατί αν δεν το καταφέρουμε δεν θα εκπληρώσουμε τις προσδοκίες των ε, πολιτών και θα αποδυναμώσουμε τελικά και τη δική μας τη θέση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πρόεδρος, θα ήθελα και εγώ να πω μερικά λόγια να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που έχουν ε, σχέση και με τις δικές μου τις ε, τροπολογίες. Καταρχήν, βεβαίως είχαμε τη συναπόφαση για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό βέβαια ε, είναι κάτι καινούριο για μας, ε, είναι μετά τη Λισαβόνα. Τώρα βρισκόμαστε λοιπόν σε νέα δεδομένα και το, κοινοβούλιο, συγγνώμη, το Συμβούλιο πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχουμε και εμεί φωνή, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαμε. Η Επιτροπή λοιπόν αυτή προσπάθησε να ε, δρομολογήσει την τριμερή συζήτηση, όχι με την επιτυχία που θα θέλαμε. Διαπίστωσα ότι μερικά από αυτά που λέμε εμείς ε, επικαλύπτονται με αυτά που λέει η Επιτροπή Κρίσης. Εμείς όμως, είμαστε η Νομοθετική Επιτροπή, γι' αυτό λοιπόν είναι σκόπιμο να καταρτήσουμε μια έκθεση προνομοθετική και χαίρομαι που το κάνουμε αυτό. Δεν πιστεύω ότι πρέπει απαραίτητα να ε, συμπεριλάβουμε όλες τις απόψεις μας στην έκθεση και ούτε να περιμένουμε ότι θα υλοποιηθούν όλες μας οι προσδοκίες. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ίσως υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που δεν θα κατορθώσουμε να τα συμπεριλάβουμε στην νομοθεσία την επόμενη χρονιά, αλλά εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι πρόκειται για μια συνεχιζόμενη συζήτηση και ως εκ τούτου από τη στιγμή που θα έχουμε κερδίσει εμπιστοσύνη θα ε, αναλάβουμε και άλλα μέτρα. Γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα είναι απλά ένας κοινό παρονομαστής και τότε ίσως ε, να καταλήξουμε σε κάτι που δεν θα είναι και καθόλου φιλόδοξο. Αυτά τα γενικά μου σχόλια. Τώρα, ε, Όσον αφορά τις ε, τροπολογίες, η Βίκη αναφέρθηκε σε αυτά. Ε, ήμασταν αρκετά φιλόδοξοι. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με την Ευρωζώνη. Εγώ, εκείνο που με ενδιαφέρει είναι στους κανονισμούς να υπάρχουν εκείνα τα οποία είναι προκυκλικά απέναντι στο δημόσιο χρέος και η πίεση αυτή δεν θα φύγει αν δεν δείξουμε και εμείς τη βούληση να διορθώσουμε την κατάσταση εν ευθέτω χρόνο. Το ελάχιστο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξετάσουμε το θέμα. Και ενδιαφέρομαι για όλα αυτά διότι προκύπτουν αυτόματες συνέπειες που καθορίζουν ε, κατά πόσον μια χώρα δεν ακολουθεί το σωστό δρόμο στην ισορροπία των δαπανών. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή και το Συμβούλιο ε, παρεμβαίνουν και δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζουμε ότι και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προσπαθούν να πείσουν τις αγορές ότι όλα βαίνουν καλώς, να επιδείξουν εμπιστοσύνη για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη έτσι ώστε όλα πράγματι να πάνε καλά. Ή από την άλλη υπάρχουν εποχές όπως αυτή που ε, βιώνουμε τώρα, όπου μερικοί σιωπούν, ε, δεν θέλουμε να συζητήσουμε ε, κατά πόσον θα υπάρξουν χρεοκοπίες ή αναδιάρθρωση χρέους, γιατί αυτό θα φοβήσει τις αγορές. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σήμερα. Και το θέμα είναι τι θα γίνει μετά από δύο χρόνια εάν προκύψει μια τέτοια κατάσταση τότε η Κομισιόν θα είναι νευρική και τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, ε, να γνωρίζουμε τα πράγματα τα οποία λειτουργούν αυτόματα. Κατανοώ βέβαια ότι είναι πολύ δύσκολο ορισμένα από αυτά τα πράγματα να γίνουν βραχυπρόθεσμα, γιατί εδώ ε, μιλάμε για μηχανισμούς που προκύπτουν όταν ε, υπάρχει και κρίση. Καλό όμως τους συναδέλφους να σκεφτούν όλα αυτά και να διασφαλίσουν ότι αυτά θα υπάρχουν στην έκθεσή μας. Η ιδέα ότι είμαστε πολύ πιο διορατικοί από το να λύνουμε απλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον κοινό παρανομαστή, αυτό μακροπρόθεσμα δεν θα αντέξει στο χρόνο δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ίδιο πράγμα μετά από 10 χρόνια. Έχουμε πολύ πιο πολλή δουλειά να κάνουμε από αυτή που έχουμε μπροστά μας τώρα. Αυτά είναι τα σχόλιά μου και θα ήθελα να επανέλθω στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ξεκινώ ευχαριστώντας όλους όσοι έλαβαν το λόγο. Θέλω επίσης να ξεκινήσω απευθυνόμενος προς τον κύριο Γκίγκολντ που με πολύ έξυπνο τρόπο μου δίνει πάρα πολλές ευθύνες. Σκέφτομαι αμέσως τη συνέχιση του διαλόγου με τους σκιώδεις εισηγητές. Πιστεύω ότι στο θέμα αυτό ε, πρέπει να έχουμε ενιαία στάση. Είναι πολιτικό το ζήτημα, δεν είναι τόσο τεχνικό όσο η εποπτεία. Αλλά επιτρέψτε να πω ότι οι διάφοροι σκιώδεις εισηγητές συχνά δέχθηκαν απόψεις που δεν ήταν κατά ανάγκη δικές τους 100%. Κάποιοι προάσπιζαν περισσότερο την διακυβερνητική προσέγγιση, Άλλη τον, ε, την κοινοτική μέθοδο. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων για τον ε, ρόλο των κοινοτικών οργάνων, άλλοι είναι υπέρ της ε, πιο ομοσπονδιακής διάστασης, άλλοι αρνητικοί. Ωστόσο, όλοι οι εισηγητές έδωσαν μια θετική, είχαν μια θετική στάση προς την έκθεση και πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή κοινή θέση. Προφανώ κάποιε ομάδε είναι πιο αριστερά, κάποιε είναι πιο δεξιά. Πιστεύω ωστόσο ότι μπορούμε να έχουμε μια κοινή στάση. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για ένα τόσο λεπτό ζήτημα το να έχουμε μια ισχυρή θέση και θα προσπαθήσω με κάθε ε, μέχρι τη στιγμή της ψήφου με όλες τις δυνάμεις μου να πετύχω κάτι τέτοιο. να προσθέσω μερικά πράγματα στη, προς τον Φιλίπ και τη Σιλβία. Όντως υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν περιλαμβάνονται ε, στις συμβαστικές τροπολογίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω θετική άποψη. Δεν χρειάζεται όλες οι τροπολογίες να είναι συμβατές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα που έθεσε η η έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις βράχη και μακροπρόθεσμες. Κάποια από τα μέτρα μπορεί να απαιτήσουν στο μέλλον αλλαγή της συνθήκης. Γι' αυτό το λόγο τα μέτρα είναι διαφοροποιημένα. Κάποια μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν τώρα, άλλα απαιτούν διεξοδικότερη μελέτη. Σε ό,τι αφορά την μελέτη των μέτρων αυτών μπορούμε να αφέσουμε κάποιες προθεσμίες. Μίλησε η Ελίζα για παράδειγμα γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα να είναι σαφή τα πράγματα. Οι βασικές διαφορές αφορούν τις συστάσεις 1 και 2, ιδίως τις κυρώσεις. Δηλαδή, οι κυρώσεις θα είναι αυτόματες θα γίνονται αυτόματα ή όχι και ποιο είναι ο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Επιτροπή. Να σα πω ω προ το σημείο αυτό ότι το Κοινοβούλιο ήδη έχει ε, μια ιστορία σχετικά. Έγιναν κάποιες εκθέσεις, υιοθετούν κάποιες εκθέσεις στην Ολομέλεια, για παράδειγμα η έκθεση για την κρίση η δική μας έκθεση πρέπει να ακολουθήσει τα προγενέστερα παραδείγματα. Δεν ανησυχώ λοιπόν. Πιστεύω ότι και στο σημείο αυτό θα υπάρξει μια κοινή θέση και θέλω να πω εξ αρχής ότι ε, υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων, στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων μερικές φορές, μεταξύ βουλευτών. Το βλέπουμε άλλωστε και σε κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, διαφοροποίηση Eurogroup και υπόλοιπων κρατών της Ένωσης. Η οικονομική διακυβέρνηση είναι ιδέα για τους 27, πρέπει να έχει ωστόσο και οι ειδικέ ρυθμίσεις για το Eurogroup. Το ίδιο ισχύει και για την, ε, αυτό υπήρχε στην ε, πρόταση για την κρίση, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει και για την έκθεση τη δική μας. Σε ό,τι αφορά το, σύμφωνο σταθερότητα που είναι και ανάπτυξης, είχα πει πολλέ φορές ότι το σύμφωνο αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο και ανάπτυξη. Όταν υπάρχει ανάπτυξη της οικονομία θα έχουμε και καλύτερη θέση, καλύτερη κατάσταση της απασχόλησης. Και εδώ προτείνω να συμπεριληφθεί η ιδέα αυτή στην έκθεση. Ό,τι αφορά τώρα τα ευρωομόλογα. Έχει γίνει λόγος για το θέμα αυτό ακόμα και από τον κύριο Μπαρόζο στην Ολομέλεια του Στρασβούργο. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να μελετηθεί προσεκτικά το ζήτημα αυτό και στο μέλλον. Τελευταία παρατήρηση. Φορολογία. Το επίπεδο των δαπανών και το επίπεδο των εσόδων πρέπει να είναι βιώσιμο. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Για τα φορολογικά ζητήματα πιστεύω και εδώ υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας, ότι μπορούμε να έχουμε μια κοινή θέση, ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίες συνδιαλλαγής των διαφόρων ομάδων. Και εγώ τώρα εδώ θέλω να απευθυνθώ στους και ηγητές κυρίως, ζητώντας τους να δείξουν καλή προαίρεση για να έχουμε μια κοινή θέση. Τελευταίο ζήτημα. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι περισσότερο Κοινοβούλιο, άρα να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα ωστόσο πρέπει να είναι και περισσότερο ευρωπαϊκό. Να παίζει λοιπόν βασικό ρόλο συντονισμού με τα εθνικά κοινοβούλια. Αν έχουμε ένα κοινοβούλιο που ελέγχει καλύτερα την οικονομική διακυβέρνηση και παίζει βασικό ουσιαστικό ρόλο στις συζητήσεις για τους ε, μελλοντικούς προσανατολισμούς της Ένωσης, τότε το Κοινοβούλιο θα ανεβάσει τη σημασία του στον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι είναι δυνατό, απολύτως, έστω και οι τοπολογίες ε, κάποιων πολιτικών ομάδων είναι διαφορετικές. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει και μπορούμε να βρούμε συνένεση για το ρόλο του Κοινοβουλίου στην οικονομική διακυβέρνηση και με τρόπο ώστε να επιτρέψουμε στο Κοινοβούλιο να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο στο μέλλον. Να πω επίσης ότι ελπίζω να έχουμε μια στέρεη κοινή θέση σύντομα και να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει μια τέτοια κοινή θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι λοιπόν ε, είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα για την ε, ψηφοφορία στις 4, ε, μάλλον όχι συγγνώμη στις 5 Οκτωβρίου λέει η Πρόεδρος και θα πάμε στην τελική ψηφοφορία στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Πολύ ωραία, πάμε τώρα στο τελικό θέμα για σήμερα το οποίο είναι η πρόταση για τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις ε, που διευκολύνουν την πάυση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακοριχείων. Ο κύριος Ραπκάι είναι ο εισηγητής. Ε, θα περιμένω λίγο να έχει λίγη ησυχία. Ja, herzlichen Dank, Frau Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όταν το 2002 μετά από 50 χρόνια εξέπνευσε η ΕΚΑΧ τότε κρίθηκε απαραίτητο μεταξύ άλλων όχι μόνο για αυτό λόγο αλλά και για αυτό το λόγο να αποφασιστεί το καθεστώς κρατικών ανισχύσεων για το λιγνίτη και να εξευρεθεί μια μεταβατική διάταξη που θα μπει μέσα στη γενικότερη συμφωνία. Τότε λοιπόν υπήρξαν κανονικοί εξαιρέσεων για το λιγνίτη που είχαν διάρκεια μέχρι 31 Δεκάτου του 2010. Τότε λοιπόν υιοθετήθηκαν και οι σχετικές ρυθμίσεις από την συνθήκη της ΕΚΑΧ. Κυρίως δύο μορφές ενισχύσεων που ήταν οι ενισχύσεις για την πάυση λειτουργίας αφενός και αφετέρου οι ενισχύσεις παραγωγής. Τα λέω όλα αυτά, κυρία Πρόεδρε, διότι ένα επιχείρημα το οποίο αναφέρεται επανειλημμένα σήμερα είναι ότι τότε δεν επρόκειτο για κανονισμό πάυσης λειτουργίας. Και τότε συζητήθηκε βέβαια το θέμα αυτό, όμως σε τελική ανάλυση δεν πρόκειται για κανονισμό πάυση λειτουργίας, τότε ήταν ένας κανονισμός με συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Τότε τα οκτώ χρόνια επελέγησαν συνειδητά, διότι σύμφωνα με την τότε συζήτηση επελέγει αυτή η λύση όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικότερα για τις ενισχύσεις. Και υπήρχε μια απόφαση δικαστηρίου που έλεγε ότι οι ενισχύσεις θα πρέπει να φθήνουν και δεύτερον να έχουν και ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Ανάμεσα λοιπόν στα 5 χρόνια και τα 15 χρόνια που τότε αυτός ήταν ο χρονικός ορίζοντας συμφωνήσαμε στα 8 χρόνια διότι οι αποφάσει του δικαστηρίου κατέτειναν στο ότι το χρονικό διάστημα δεν θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο των 10 ετών. Σας το λέω λοιπόν αυτό, διότι σήμερα συζητάμε σαν επρόκειτο για ε, κανονισμό που θα εξέπνε. Εγώ τότε ήμουνα στην Οικονομική Επιτροπή ε, ήμουν πλήρες μέλος ε, και ήμουν εισηγητής για τον Λιγνίτη. Ε, μέχρι και πέρυσι ήμουν πλήρες μέλος, τώρα είμαι μόνο αναπληρωματικό. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και αν είμαι αναπληρωματικός, ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να είμαι ο εισηγητής σας για το θέμα αυτό. Το δεύτερο επιχείρημα που προβάλλεται όπως λέει και η πρόταση Κομισιόν, είναι ότι το 2014 θα εκπνεύσει οριστικά αυτό το καθεστώς και αυτό βασίζεται στην παραδοχή ότι η πάυση λειτουργίας ε, εκμετάλλευση λιθάνθρακα με ενισχύσει στην Ευρώπη, το γεγονός αυτό θα συνέβαλε στη βελτίωση των κλιματικών συνθήκων. Αυτό όμως δεν είναι εύκολα κατανοητό, διότι καταρχήν η ο εγχώριος άνθρακας θα αντικατασταθεί με εισαγόμενο άνθρακα και κατά δεύτερον εδώ πρόκειται μόνο για τον επιδοτούμενο άνθρακα. Υπάρχουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές εξορίξεις άνθρακα χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς ενισχύσεις, οι οποίες αυτές εξορίξεις δεν αγγίζονται καθόλου. Ένα άλλο τρίτο θέμα που θέλω να αναφέρω ότι βέβαια μπορούμε να διαφωνήσουμε γι' αυτό, αλλά κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, ε, είναι κατά των ενισχύσεων για λόγους αρχής. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η συνθήκη ξεκινάει από την απαγόρευση ενισχύσεων, αναφέρει όμως ότι μπορούν να υπάρχουν και εξαιρετικές συνθήκες και αυτή εδώ θεωρείται μια εξαιρετική περίπτωση. Και αυτό πάλι το λέω διότι η Επιτροπή με την πρότασή της που λέει ότι όλα αυτά θα εκπνεύσουν το 2014, κατά τη δική μου άποψη η Κομισιόν καταθέτει μία πρόταση έολη, παντελώς έολη. Τουλάχιστον ε, η αξιολόγηση επιπτώσεων της ε, Κομισιόν δεν αναφέρει κανένα λόγο. Εγώ σας ανέφερα κάποιους λόγους, αλλά όλοι αυτοί ε, στην αξιολόγηση επιπτώσεων απαντώνται με τον τρόπο που σας παρουσίασα, άρα δηλαδή δικαιολογείται κανείς να ισχυριστεί ότι το 2014 η τελική ημερομηνία εκπνοής, που δεν είναι καν τέσσερα χρόνια, γιατί η εκπνοή του κανονισμού θα είναι κατά τα μέσα του 2014 και όχι κατά το τέλος. Αυτή λοιπόν η προθεσμία είναι αυθαίρετη. Όλα τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην αξιολόγηση επιπτώσεων, όλα αυτά βασίζονται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όχι σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, αλλά σε μεγαλύτερο. Παραδείγματο χάρη το γεγονό ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν είναι πια πολλά όπου να ε, φλέγει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν όμως κάποια που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές των κρατών μελών. Το 2014 ε, σε ορισμένα κρατημέλια αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν μεγάλες κοινωνικές αναταραχές, ότι θα υπάρξουν απολύσει, ότι θα κλείσουν εργοστάσια και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Γερμανία, αλλά ισχύει και για την Ισπανία και για τη Ρουμανία και ίσως ισχύει και για άλλες χώρες. Εκείνο το οποίο είναι εκνευριστικό είναι το γεγονός ότι η Κομισιόν έχει κάνει μια πολύ καλή αξιολόγηση επιπτώσεων. Μόνο που στην απόφαση της ε, στο σώμα των επιτρόπων δεν τηρεί αυτή την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Ο συνάδελφος κύριος Αλμούνια αναφέρει μια άλλη ημερομηνία που είναι πολύ πιο κοντά από αυτήν που αναφέρεται στην ε, πρόθεση Κομισιόν. Ο κύριος Αλμούνια αναφέρεται στο 2018 και αυτή η ημερομηνία προκύπτει από το εξή σκεπτικό. Υποτίθεται εκπνέει ο κανονισμό. Θα πρέπει όμως να υπάρχει ικανοποιητικό χρονικό διάστημα έτσι ώστε κλιμακούμενα να ε, καταργούνται οι ενισχύσεις με φθήνουσα πορεία έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των ε, κοινωνικών ανταρχών. Γιατί εάν ε, η ημερομηνία είναι πολύ πιο κοντά, τότε θα υπάρξουν πράγματι μεγάλα προβλήματα. Εγώ λοιπόν θεωρώ και αυτό αναφέρω στην ε, έκθεσή μου ότι η ημερομηνία της 1ης Οκτωβρίου του 2014 να μετατεθεί στην 31η Δεκάτου του 2018. Εδώ πρέπει να ληφθούν και κάποια άλλα τεχνικής φύσεως μέτρα. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι η πρόταση της Κομισιόν αγνοεί παντελώς ε, τα συμπεράσματα της αξιολόγησης επιπτώσεων. Αν πραγματικά τηρηθεί η ημερομηνία 2014, μιλάμε για 45 μήνες, 3 επί 15 δηλαδή, 3 επί 15 μήνες, άρα 33% μείωση των ενισχύσεων σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι πρόβλημα. Αντί για 33% αν παίρναμε το 15% θα φτάναμε στο 101% και αυτό δεν γίνεται μαθηματικά. Η Κομισιόν λοιπόν δεν κατορθώνει με τις ε, ρυθμίσεις της να αναστείλει τους νόμους της μαθηματικής. Και αυτό το 33% είναι ανόητο. Παρ' όλα αυτά σας λέω πρέπει να είναι ε, κλιμακούμενη προς τα κάτω η μείωση των ενισχύσεων. Γι' αυτό εγώ μιλάω για 8 χρόνια. Με ένα 10% τουλάχιστον, εδώ ταιριάζει το τουλάχιστον, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να κατανοήσει ότι ε, κάποιες χρονιές μπορεί να υπάρξει και ταχύτερη ε, περικοπή των ενισχύσεων. Πάντως εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ πιο αποδεκτό ε, σε επίπεδο κοινωνικών ταραχών. Υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις στην πρόταση Κομισιόν όπου εγώ δεν διαφωνώ του Ναντίον θα τις υποστήριζα, μόνο που εδώ βέβαια ε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί δεν έχουν σχέση με την ουσία. Παραδείγματο χάρη, σε σχέση με τα ε, προγράμματα παύσης ε, λειτουργίας, αναφέρονται και περιβαλλοντικά προγράμματα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, μόνο που αυτό θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο του άνθρακα γιατί να ισχύει, μόνο για τον λιθάνθρακα. Έχουμε σε κάποια κράτη-μέλη που εξάγονται ακόμα μεγαλύτερες ε, ποσότητες ε, και εκεί δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω λοιπόν ότι το αίτημα ε, σε επίπεδο αρχή είναι σωστό, όμως θα πρέπει να ρυθμιστεί το πρόβλημα μέσα από σχετική νομοθεσία. Δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί το θέμα μέσα από έναν κανονισμό απαλλαγή. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές ε, οι απόψεις μου που περιλαμβάνονται στο σχέδιό μου και ανακεφαλαιώνω πρώτον να υπάρξει παράταση μέχρι το 2018 ε, σε, σε σχέση με αυτό τον κανονισμό που εκπνέει τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι μετά το 2018 γενικά θα καταργηθούν οι ενισχύσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, έχω καταθέσει δύο τροπολογίες όπου αναφέρω την πρόταση να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε ανταγωνιστικός και μη ανταγωνιστικός. Διότι οι εγκαταστάσεις εκείνες οι οποίες Αυτό εξάλλου και το σκεπτικό των ενισχύσεων, να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα. Εάν ευθύ εξ αρχής κλείσουν όλες οι εγκαταστάσεις, ακόμα και εκείνες που θα μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικές, αυτό δεν το βρίσκω σωστό. Γι' αυτό λοιπόν προβαίνω σε αυτό το διαχωρισμό σε ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές ε, εγκαταστάσεις. Επίσης, ε, από τον ισχύοντα κανονισμό ε, πήρα τρία, τρεις σκέψεις ε, και θα ήθελα να τις συζητήσουμε, οι οποίες ε, σκέψεις αυτές ε, συμβαδίζουν και είναι στο πνεύμα της αξιολόγησης επιπτώσεων. όπως παραδείγματος χάρη και κάποιες σκέψεις που αναφέρονται στην πρόταση Κομισιόν. Όλα αυτά, αν θέλετε, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Όσον αφορά τώρα στο χρονοδιάγραμμα, το αργότερο το Νοέμβρη πρέπει να πάμε στην Ολομέλεια, διότι νομίζω στις 10 ε, Δεκεμβρίου θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνισμού. Το θέμα είναι ότι εκείνοι που δεν επιθυμούν ε, καθόλου στις ενισχύσεις ε, εδώ πρέπει να πούμε ότι μέχρι το τέλος του κανονισμού πρέπει να υπάρχει ένας νέος κανονισμός. Αν δεν υπάρχει κανονισμός δεν ισχύει ούτε το 2014. Και με βάση τη συνθήκη 1η του 2011 οποιαδήποτε μορφή ενίσχυσης ε, παραβιάζει τους ε, κανονισμούς. Άρα δηλαδή ε, για να ισχύσει το αντίθετο θα πρέπει να δοθεί έγκριση κομισιών και αυτό είναι πολύ πιο αυστηρό ε, παρά από τον να ε, ισχύει ο κανονισμός ε, για συγκεκριμένο τομέα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι μέχρι τον Νοέμβρη πρέπει να έχει κλείσει το θέμα, άρα δηλαδή αρχές Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουμε ψηφίσει στην Επιτροπή μας και από εκεί θα προκύψουν οι υπόλοιπε γραμματείε, τι οποίε τι ε, υπόλοιπε ημερομηνίες τις οποίες γνωρίζει η γραμματεία. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση στις 9 Νοεμβρίου να ψηφίσουμε. Αρχικά είχε προβλεφθεί την επόμενη εβδομάδα να γίνει συζήτηση, του όμως ε, λόγω της ημερήσιας διάταξης δεν γίνεται, στη ημερήσια διάταξη επόμενης εβδομάδας, άρα δηλαδή θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση ε, όσον αφορά στις τροπολογίες. Πάντως, σε επίπεδο αρχής, νομίζω ότι μπορούμε να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Όπως ε, μίλησε για το χρονοδιάγραμμα ο, προ, ο εισηγητής, θα ήθελα να πω ότι πράγματα υπάρχει κατάθεση της πρώτης πρότασης 5 Οκτωβρίου, 11 Οκτωβρίου η κατάθεση των τροπολογιών, συζήτηση 26 Οκτωβρίου, ψηφοφορία 9 Νοεμβρίου και ελπίζω να είμαστε στην Ολομέλεια την δεύτερη του μηνός Νοεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας. Κύριε Λάγκεν, έχετε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, εδώ το θέμα δεν είναι να χορηγούνται ευρωπαϊκές ενισχύσεις, αλλά εδώ πρόκειται για την χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Βασικά ο συνάδελφος κ. Ράπκαη σωστά είπε ότι οι εναλλακτικές λύσεις που αναζήτησε η Κομισιόν είναι έξι και αυτές ε, δεν συμβαδίζουν, έχουν καμία σχέση με τον κανονισμό. Η Κομισιόν αναφέρθηκε σε μια εναλλακτική πρόταση υπαριθμών 5 η οποία εγγυάται ένα δεκαετές πρόγραμμα για την πάυση λειτουργίας των ε, ε, καταστάσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κατά την Κομισιόν αυτή είναι η βέλτιστη λύση. Μετά όμως, ξέρουμε πώς προέκυψε αυτή η λύση, αποφασίστηκε στο Σώμα των Επιτρόπων. Ε, το 2018 ε, δεν υπερψηφίστηκε και γι' αυτό η Κομισιόν προτείνει το 2014. Αυτό λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με τις εναλλακτικέ άλλες λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κοινωνική διάσταση του θέματος και τη συνθήκη. Ο κύριος Ράπκαϊ το έκανε αυτό, ε, κατέθεσε ένα σχέδιο που δεν έχει όμως ακόμα μεταφραστεί, βρίσκεται τώρα στη μετάφραση, παρουσίασε εν πάση περιπτώσει τις απόψεις του και εγώ πιστεύω ότι το ερώτημα πώς μπορούμε 100.000 θέσει εργασία σε τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπιστούν και ε, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε μια ήπια εκπνοή της χορήγησης ενισχύσεων, αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα στον κανονισμό ε, περί διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί αν δεν υπάρχει πλέον εξόριξη εγχώριου άνθρακα και αυτό αυτός ο άνθρακας ενισχύεται γιατί δεν είναι ανταγωνιστικός, τότε προφανώς θα εισάγεται άνθρακας. Ε, το διοξείδιο του άνθρακα δεν μπορεί να είναι ε, η αιτιολογία, η πολιτική για διοξείδιο του άνθρακα, τη στιγμή που συμφωνούμε όλοι ότι ε, θα πρέπει να εμπλωτιστούν υπάρχουν υπάρχουσες μορφές ενέργειας και υπάρχουν συνολικά 12 πιλωτικά προγράμματα. Εγώ ως μέλος ε, της Επιτροπής Βιομηχανίας το γνωρίζω αυτό. Υπάρχουν 12 προγράμματα για την δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτά πηγαίνουν παράλληλα. Υπάρχει σαφώς ε, ενασχόληση με τα θέματα τα περιβαλλοντικά. Εδώ τι το ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριος Ραπκάι λέει παράταση μέχρι το 18, αντί για το 14. Στη Γερμανία αυτό από το 2007 είναι νόμος. Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει σύμπτωση. Βεβαίως η Κομισιόν μόνη της παρουσίασε την αλλακτική λύση 6, η οποία λύση αυτή λέει ότι μπορεί να υπάρξει παράταση για άλλα 10 χρόνια και μετά να υπάρξει πλήρης πάυση ε, των ενισχύσεων. Ε, μπορεί κανείς να τα ζυγίσει αυτά τα δύο. Το πιο λογικό θα ήταν, και το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια, το πιο λογικό λοιπόν θα ήταν η Κομισιόν να αποσύρει την πρότασή της για το 2014 και να επανέλθει στην παλιά πρόταση του κ. Αλμούνια για το 2018. Και αν το έκανε αυτό η Κομισιόν θα μπορούσε να τύχει εδώ η πρόταση Κομισιόν ευρεία συνένεση. Ε, μάλιστα αυτό το πρότεινε ο Υπουργό Αρμόδιος ε, για τα θέματα βιομηχανία. Και θα μπορούσε λοιπόν να ξεβρεθεί μια λογική κοινωνική λύση. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Εγώ ελπίζω η Κομισιόν να αντιμετωπίζει αυτήν την κατάσταση. Ο αρμόδιος ε, επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού καταψηφίστηκε. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να διορθώσει η Κομισιόν το λάθος της και κατά τα άλλα ε, υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την πρόταση του αδέλφου κυρίου Ράπκαη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Δεν είμαστε κατά των επιδοτήσεων αυτών. Αυτό το θέμα, το, το μέσο βέβαια μας απασχόλησε γιατί μερικές φορές χρηματοδοτεί ε, βιομηχανίες οι οποίες μολύνουν την ατμόσφαιρα. Το θέμα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι ότι υπάρχουν εδώ δημόσια χρήματα που δίδονται προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά δεν πρέπει να δαπανηθούν δύο φορές, αλλά μόνο μία. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι η οικονομική τους αποτελεσματικότητα πώς εμείς μπορούμε να διασφαλίσουμε διαρκείς θέσεις απασχόλησης στο σύνολο της Υπήρου χρησιμοποιώντας τα χρήματα αυτά. Έχουμε δει ότι τα ίδια και με την αυτοκινητοβιομηχανία. Έχουμε διαθέσει δισεκατομμύρια προς τη βιομηχανία αυτή χωρίς προϋποθέσεις και αυτό που βλέπουμε είναι ότι ε, στις νέες χώρες επενδύουν ε, οι επιχειρήσεις αυτές ε, και επενδύουν και οι νέες αυτές χώρες σε νέες τεχνολογίες και εμείς δίνουμε λεφτά σε βιομηχανίες οι οποίες ξέρουμε ότι θα διαφύγουν και τα συζητούσαμε αυτά με τον Τρισέ. Το θέμα λοιπόν είναι να διασφαλίσουμε την οικονομική αποδοτικότητα των χρημάτων ε, τα οποία δαπανάμε προς την κατεύθυνση αυτή γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι δεν γίνεται σωστή χρήση. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να δώσουμε τα λεφτά αυτά, θέλουμε όμως τα λεφτά αυτά να πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Και εδώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλοδεχούμενη. Να πούμε ότι φεύγουμε από την ε, κατεύθυνση αυτή και επιταχύνουμε την καινοτομία και τις επενδύσεις σε ε, βιομηχανίες με μέλλον. Λυπάμαι γιατί πρέπει να φύγω πια και δεν θα ακούσω αυτά τα οποία θα πει ο εισηγητής. Αλλά τις επόμενες μέρες θα μας δοθεί η δυνατότητα συζήτησης. Έτσι και αλλιώς πέντε λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, Σίμων. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως να προλάβετε να ακούσετε τι θα πω. Νομίζω ότι όλοι εδώ συμφωνούμε ότι ε, θέλουμε πιο ενέργειες πιο φιλικές προς το περιβάλλον και συμφωνούμε όλοι ότι ο δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των κρατικών δαπανών. Ο κύριος Λάγκεν πολύ σωστά είπε ότι εδώ δεν είναι κοινοτικά τα κονδύλια, εθνικά είναι. Και έρχομαι λοιπόν εγώ από την Επιτροπή ε, Περιφέρειας, Περιφερειών και ε, εκεί γίνεται λόγος πώς θα δαπανώνει τα χρήματα στο μέλλον. Εδώ λοιπόν έχουμε μία μακροπρόθεσμη προοπτική. Αν την χάσουμε αυτή και αν χάσουμε και την κοινωνική διάσταση, αν ε, χάσουμε την οπτική γωνία των θέσεων εργασίας, τότε δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γιατί φτάνουμε στο ερώτημα τι θα γίνει με τα εθνικά κονδύλια, με τα κοινοτικά κονδύλια και ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Ράπκαη το είπε και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Υπάρχει στην πρόταση του κύριου Ράπκαη ε, το να υπάρχει ένα κατώτατο όριο και νομίζω και εδώ και σε άλλες επιτροπές όταν μιλάμε για τεχνολογικό άλμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν λέμε ότι θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι στην τεχνολογία να έχουμε κατά νου ότι όσον αφορά στην εξόριξη του άνθρακα είμαστε πρωτοπόροι και για να διατηρήσουμε τη θέση μας ε, πρέπει και στο μέλλον να διασφαλίσουμε την επιβίωση του τομέα γιατί αν δεν έχουμε εμείς ε, τα δικά μας τα λιγνητορυχεία, θα υπάρχουν αλλού. Το μόνο που θα κάνουμε εμείς είναι θα συμβάλλουμε εμείς τα δικά τους να είναι πιο οικολογικά. Πρόεδρος. Τα κακά νέα είναι και εγώ πρέπει να φύγω. Άρα όντως το και μισή θα κλείσουμε. Ο κύριος Νίτρα ζήτησε το λόγο. Και με δύο λόγια θα τα πω, Πρόεδρε, για να φύγετε. Συμφωνώ με τον κύριο Λάγκες που έφυγε και αυτός. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την διακοπή λειτουργίας ε, ανθρακοριχείων που δεν είναι οικονομικά αποδε, ε, οικονομικά βιώσιμα, διότι ε, η κοινωνία θα πρέπει να... δεν μπορεί να πληρώνει εσαΐ το κόστος. Καταλαβαίνω τον κύριο Λάγκεν που λέει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ε, κάτι τέτοιο στα, στα κυβερνητικά προγράμματα. Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα με την κάλυψη των έκτακτων ε, δαπανών. Δεν διάβασα το κείμενο στα αγγλικά μέχρι τώρα, μόνο στα γερμανικά υπάρχει. Λυπούμε γι' αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Ε, και να διατηρηθώ αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε. Είπατε, τουλάχιστον έτσι κατάλαβα, ότι στο άρθρο 3 Β, το άρθρο 3 Β να καταργηθεί. Δηλαδή, η βοήθεια, ανεξάρτητα από την ημερομηνία, πρέπει να δίδεται στη, στα αρθρακοριχεία που ε, κλείνουν. Εάν φύγει η παράγραφος αυτή, σημαίνει ότι η βοήθεια αυτή ε, θα πρέπει να δοθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά γιατί μιλάμε για την χρηματοδότηση του κλεισίματος ή την χρηματοδότηση των ανθρακοριχείων. Να δώσω το λόγο το ξανά στον εισηγητή. Έχει δύο λεπτά. Ξέρετε, δεν πάω σε κοκτέιλ και άλλες δουλειές έχω, οπότε μην με κατηγορείτε. Ζητώ συγγνώμη από του άλλου ομιλητέ, αλλά πρέπει να κλείσουμε ακριβώ την ώρα μα. Κύριε Ράπκαη, μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα του κύριου Νίτρος. Ούτω ή άλλω, ε, πρώτη ανταλλαγή από όποιον κάνουμε σήμερα. Όταν δούμε το κείμενο θα μπορέσουμε να ξαναζητήσουμε το θέμα. Κύριε Ράπκαη. Κοιτάξτε, λέω από συναδέλφου ότι εγώ δεν προτείνω να διαγράψουμε το άρθρο 3α, κάθε άλλο. 3α ή 3β λέει ο μιλητής. Υπάρχει ε, το 3 παράγραφος α ή παράγραφος β. Εγώ δεν θέλω να διαγραφεί καμία τύπο, παράγραφος τίποτα. Εγώ ε, θέλω μόνο ε, να αλλάξει ημερομηνία. Και κατά τα άλλα επισημαίνω ότι χρειαζόμαστε το πρόγραμμα πάυσης λειτουργίας εφόσον τα εργοστάσια ή τα ανθρακοριχεία δεν είναι ανταγωνιστικά δεν θέλουμε να χορηγούμε ενισχύσεις σε κάτι που δεν χρειάζεται πλέον ενισχύσεις. Εγώ το μόνο που θέλω να καταστήσω σαφές είναι ότι θα ήθελα να συζητήσω με τους ε, συναδέλφους ε, διότι ο συνάδελφος που μόλις τώρα έφυγε κάνει ένα θεμελιώδες λάθος. Λέει ότι ο άνθρακας είναι ξεπερασμένος. Μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά υπάρχει και σήμερα και θα υπάρχει και αύριο. Και ο συνάδελφος κύριος Σίμων το επισήμανε. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως ο λιθάνθρακας θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία ανά τον κόσμο. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο και το αέριο, ε, ο λιθάνθρακας ε, έχει τεράστια αποθέματα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το εξετάσει κανείς και από πλευράς τεχνολογικής και από πλευράς υπεραξίας. Εγώ συνάδελφε δεν διέγραψα τίποτα, απλά ε, για λόγους καθαραλογικούς, αλλάζω την ημερομηνία. Ο συνάδελφος κύριος Λάγκεν μίλησε για 10 χρόνια και εγώ αρχικά 10 χρόνια είχα να προτείνω, μου θύμισε όμως την παλιά κουβέντα που είχαμε κάνει και όπου είχαμε πει να μην είναι διψήφιο ε, διψήφιος αριθμός. Ο κύριος Αλμούνια ο ίδιος και το τονίζω, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έκανε πολύ καλή δουλειά στην περίπτωση αυτή. Ε, οι άλλοι επίτροποι δεν τα κατάλαβαν. Εγώ λοιπόν είπα 2018 με βάση αυτό το σκεπτικό να υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας και με βάση το ότι ο ίδιος ο Επίτροπος πρότεινε συνεδρίες της Επιτροπής το 2018. Γι' αυτό λέω και εγώ 18. Αρχικά είχα πει και εγώ 2020. Τέλο πάντων, να το κουβεντιάσουμε αυτό. Ε, γνωρίζω από την ε, Επιτροπή Περιφερειών ότι εκείνοι πρότειναν το 2020, το είπε και ο κύριο Ζήμων, που έρθει από την Επιτροπή, θα το συζητήσουμε. Sorry, is somebody calling for the floor? Κάποιος είπε κάτι. Ξέρω ότι δεν μιλήσατε και άλλοι δεν μιλήσανε, αλλά δεν έχουμε χρόνο, θα έχουμε άλλες ευκαιρίες. Λοιπόν, διακόπτουμε εσάβριον.